ladies Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την απογευματινή μας ε, συνεδρίαση αμέσως με μεγάλη χαρά. Έχουμε μαζί μας και καλωσορίζω τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας ε, της ΚΝΕΣΕΤ, τον κύριο Τζάκι Χανέγκμπι. είναι λίγο δύσκολο να προσφέρω το όνομά σας. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητέ ε, κύριε Χανέκμπη, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας ε, που είναι η ε, Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνα του Κοινοβουλίου. Θέλουμε να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας και τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε μαζί σας σήμερα αφορούν τις παγκόσμιες απειλές κατά της ασφάλειας, καθώς επίσης και ιδιαίτερως οι επιπτώσεις τους στην Μέση Ανατολή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θέλουμε λοιπόν κάποιες, ε, δεν θέλουμε τη δικιά σας άποψη ε, όσον αφορά τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τη δικιά σας άποψη για τα τεκτενόμενα από τη μεριά της Μέσης Ανατολής. Ο Πρόεδρο ε, τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνα τη Κνεσέτ, ο κ. Χανέγκμπι, ήταν ήδη χθε ε, καλεσμένος τη επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, τη ΑΦΕΤ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά εμείς εδώ ε, θα εστιάσουμε την προσοχή μας περισσότερο σε απειλές κατά της ασφάλειας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Το ε, Ισραήλ είναι φίλος και συνεργαζόμενο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν αμέσως θα σας δώσω το λόγο χωρίς να καθυστερήσω άλλο obtain your reflections. The is yours. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της ε, Υποεπιτροπής ε, Ασφάλειας ε, και Άμυνας του Κοινοβουλίου. Είμαι εδώ μαζί με κάποιους συναδέλφους μου, τους οποίους θα σας παρουσιάσω σύντοση λίγο. Προσεκλήθημεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Είχαμε μια σειρά επαφών με διάφορους φορείς. Χθες ε, συναντηθήκαμε με πολλά σημαντικά άτομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όπως είπατε, είμαστε καλεσμένοι και στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής ΑΦΕΤ και του Προέδρου κ. Μπρόκ, με τον οποίο αργότερα ε, ε, είχαμε και περαιτέρω συνάντηση και με την υπερτή ε, εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνη, επίσης τον Υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου, αύριο με τον αντίστοιχο Υπουργό της, των Κάτω Χωρών, τον Υπουργό δηλαδή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και είμαστε σήμερα και εδώ γιατί ε, ακριβώς ε, η φύση της δικής μας ε, Επιτροπής έχει ένα μεγάλο σκέλος για άμυνα και ασφάλεια γιατί καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς είναι από τα μεγαλύτερα μελήματα της χώρας μου και οι Υπηρεσία πληροφοριών και ο στρατός, οι Υπηρεσία ασφάλειας ε, η Μοσάντ ε, καθώς επίσης και οποιοδήποτε, ε, οποιαδήποτε διάσταση του κυβερνοχώρου που μπορεί να έχει σχέση με την ασφάλεια είναι ακριβώς εμπίπτη στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της ΚΝΕΣΕΤ. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την αντιπροσωπεία μας. Έχουμε μαζί μας τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ο οποίος ε, με μεγάλο επαγγελματισμό φέρει σε πέρα στα καθήκοντά του. Είναι από τους πιο σημαντικούς μας διπλωμάτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη που είσαστε μαζί μας και μας συνοδεύετε. Έχουμε τρία μέλη του Κοινοβουλίου από, διαφορετικές πολιτικές, ε, ε, από διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Είμαστε τέσσερι εκπρόσωποι διαφορετικών κομμάτων. Δύο από την ε, κυβέρνηση, δύο από την αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να έχουμε διεθνή αποστολή παρά μόνο εάν είμαστε, αν έχουμε ισομερή εκπροσώπηση της κυβέρνησης, της συμμαχίας κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Ε, είμαστε σαν τον Μπόλεκ και τον Λόλεκ. So, my friend from the opposition. Έχουμε τους φίλους λοιπόν από την αντιπολίτευση. Ο Εράς Μιχαήλη. Ή, συγγνώμη. Είναι η δεύτερη φορά που εκλέγεται στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Είναι έγκριτη εκπρόσωπος ε, το, του Εργατικού Κόμματος και όταν είμαι εδώ μαζί της Ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά ε, στη, στο Ισραήλ. Έχουμε τον ε, κύριο Ιάκο Πέρι, ε, τέος Υπουργό για την Επιστήμης και Τεχνολογίας. και 32 χρόνια ήταν επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας του ε, Ισραήλ και τώρα είναι επικεφαλής της ε, Υπηρεσίας. Είναι επίσης εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Λαπίντ που ήταν Υπουργός ε, Οικονομικών στην προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε τον Μάικ Ρόρετ. ο οποίος ε, ε, ήταν για χρόνια ε, υψηλός μας εκπρόσωπος στη, στην Ουάσιγκτον. Ήταν αυτός που προετοίμασε την συνάντηση Νετανιάχου Ομπάμα και αυτός που διασφάλιζε την συνέχιση των καλών σχέσεων του Ισραήλ με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Έχει γράψει πολλά βιβλία για την ασφάλεια και την πολιτική και είναι μέλος ε, της ε, Κουλάνο. Ε, της οποίας μέλος είναι και ο κύριος Μωσέ Καχλών, ο οποίος είναι ο τωρινός Υπουργός Οικονομικών. Εγώ δε εκπροσωπώ το Λικούντ. Νομίζω ότι λαμβάνοντας υπόψη ε, και την ε, ε, κατάσταση νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να ακούσουμε τα ερωτήματα μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε γιατί θα θέλαμε να έχουμε διάλογο και να ακούσουμε περισσότερο τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα των μελών της Επιτροπής σας. Εντάξει, εντάξει λέει η Πρόεδρος, γιατί όχι. Πρώτα απ' όλα, ο πρώην ε, πρόεδρος της Επιτροπής ε, ΣΕΝΤΕ, Ασφάλειας και Άμυνας δηλαδή, ο κύριος Δονζό. Εγώ θα είμαι η τελευταία που θα υποβάλω ερωτήσεις. Ε, θα ακουστώ κι εγώ, μην νομίζετε ότι δεν θα πω την απόψή μου. Ο κύριος Δονζό, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της ΚΝΕΣΕΝΤΕ. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ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 κύριε Πρόεδρε, ε, ότι θα είχα πάρα πολλές ερωτήσεις να σας υποβάλω φυσικά. Ε, και μια και εσείς δεν κάνατε μια ε, πρώτη παρουσίαση, θα μπω απευθεία στην ουσία του πράγματος. Ξέρετε ότι για μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόλυτη προτεραιότητα στη Μέση Ανατολή Έχουμε ένα πρόβλημα με την μετάφραση. Τα ακουστικά του κυρίου Χανέγκμπι δεν λειτουργούν. Έλεγα λοιπόν ότι η προτεραιότητά μας στη Μέση Ανατολή είναι βεβαίως οι σειράξεις στο Ιράκ και στη Συρία, ιδιαίτερος δε η ε, μάχη κατά ε, του ε, ISIS. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, μπορούμε να καταλάβουμε ότι, το, ε, ότι αυτό δεν είναι η στρατηγική προτεραιότητα του κράτους του Ισραήλ που έχει πιο, άμεσες, ε, πιο άμεσους ε, προβληματισμούς σχετικά με την ασφάλεια. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς αυτήν την απειλή που είναι βεβαίως απειλή αυξανόμενη στα σύνορά σας. μία απειλή η οποία σχετίζεται ε, και με την ε, Παλαιστίνη γιατί γίνεται όλο και περισσότερο λόγος ε, για την προέλευση τζιχαδιστών ε, από, τις ε, χώρες, από την χώρα αυτή, από την Παλαιστίνη και επίσης ε, το, ο Λίβανος και η Ιορδανία έχουν ήδη τοποθετηθεί απέναντι στο θέμα αυτό. Μήπως λοιπόν θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για τις δράσεις τις οποίες θα μπορούσε να αναλάβει το κράτος του Ισραήλ άμεσες ενδεχομένως, αλλά κυρίως τις δράσεις συνεργασίας που θα μπορούσε το Ισραήλ να έχει με ορισμένες από τις γειτονικές χώρες έτσι ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση αυτής ε, της απειλής του Ισλαμικού κράτους. Δεύτερη ερώτηση. Βλέπουμε καθαρά στην ε, σύραξη της ε, Συρίας ότι το Ιράν φαίνεται να ε, ε, ε, να παίζει μεγάλο ρόλο. Πώς το βλέπετε αυτό όσον αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στο περιβάλλον σας. Αναφέρομαι κυρίως στον ρόλο που παίζει σε αυτήν την ενδυνάμωση της κατάστασης που, το ρόλο μάλλον που παίζουν οι Λιβανέζοι, η Χεσμολά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Chair, Mr. Henry. Πίτσουλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ε, βλέπω ξανά. Ε, είχαμε ειδωθεί τελευταία φορά 1,5 χρόνο πριν όταν ε, η αποστολή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είχαν επισκεφθεί την ΚΝΕΣΕΤ και τότε είχαμε συζητήσει θέματα σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια. Δράτω της ευκαιρίας που μου δίδεται για να σας, να σας κάνω μια ερώτηση σε σχέση με κάτι που αναφέρατε εσείς και οι συνάδελφοι σας στην ΚΝΕΣΕΤ. Ήταν σχετικά με τις ε, ε, περίπλοκες σχέσεις με την Τουρκία. Τότε ε, αναφέρθηκε ότι υπήρχαν κάποιες ε, δυνατότητες βελτίωσης των σχέσεων με την ε, Τουρκία. Αυτό το λέγαμε 1,5 χρόνο πριν. Εν τω μεταξύ όμως ε, βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι η Τουρκία έγινε πλέον σημαντικός παίχτης στα πλαίσια της προσφυγικής κρίσης και λόγω της ροής της μεγάλης των προσφύγων που περνούν από την Τουρκία. Με ποιο τρόπο βλέπετε εσείς τον ρόλο της Τουρκίας στην Μέση Ανατολή και βεβαίως θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω και την άποψή σας όσον αφορά την ε, ανάμειξη της ε, Ρωσίας, αυτό το τρίγωνο ας πούμε Ρωσία, Τουρκία, Ισραήλ γιατί και εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, στην άμεση γειτονιά σας τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Ε, είναι πολύ περίπλοκα και ένα πράγμα που είναι δύσκολο είναι η Αίγυπτος, ε, το Σινά που είναι πολύ κοντά σας, στην γειτονιά σας. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά με την κατάσταση στο όρος Σινά. Αυτό το κομμάτι της ε, Χερσονήσου. Δεν ξέρω κάτω από ποιο έλεγχο βρίσκεται. Μοιάζει να μην είναι υπό απόλυτο έλεγχο και υπάρχει κίνδυνο και για τους κατοίκους και για τους τουρίστες σε αυτή την περιοχή. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη έχει σχέση με το Ιράν. Μετά αυτή την ε, συμφωνία για τα πυρηνικά ανάμεσα στο Ιράν και σε διάφορες χώρες βλέπετε να έχει αλλάξει η κατάσταση. Και τι γίνεται με την άρση κάποιες, ε, κάποιων από τις κυρώσεις. Θεωρείτε ότι θα υπάρξουν ε, αρνητικές εξελίξεις για την ασφάλεια του Ισραήλ ή βλέπετε να υπάρχουν ίσως και κάποιες θετικέ εξελίξεις ότι κάτι που μπορεί να αλλάξει λόγω αυτής της συμφωνίας στη σχέση σας με το Ιράν. Ευχαριστούμε κύριος Μάικλ Γκάλα. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζουμε, ε, είπε ο κ. Γκάλερ και στα εβραϊκά, καλωσορίζουμε την ε, αντιπροσωπεία από την Κνεσέτ. Το θέμα είναι ότι μπορεί κανείς να ακούσει πολλές απόψεις κυρίω στην περίπτωση τη δική σας που έρχεστε από το Ισραήλ, γιατί και εσείς στο Ισραήλ έχετε τόσο διαφορετικές απόψεις για ορισμένα θέματα, όσο και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Άρα η ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους τη ΚΝΕΣΕΤ είναι πάντα ιδιαίτερα επικοδομητική. Ε, με όσου δεν ε, είναι πλέον αξιωματούχοι και έχουν κατ' ουσίαν κλείσει το επαγγελματικό σκέλος της ζωής τους έχω διαπιστώσει ότι με όλους αυτούς συμφωνώ πολύ καλύτερα από ότι με άλλους ε, που κατέχουν πολιτικά αξιώματα. Αυτά εν είδη ε, παράπλευρης παρατήρησης. Τώρα, μία ερώτηση. Αυτό το θέμα της ε, πολυμορφίας και των πολυεπίπεδων προβλημάτων στη Συρία πώς ακριβώς τα αξιολογείτε, κυρίως έχοντας κατά νου τα σύνορα τα οποία εσείς έχετε αναλάβει να φυλάσετε. Βλέπουμε ότι από τη μια μέχρι το 2011 είχατε βρει ένα modus vivendi με τον Ασάντ, ένα τρόπο να συμβιώνετε μαζί του. Τα σύνορα ήταν ήρεμα, είχατε πρόβλημα παλαιότερα ε, για τη διέλευση της Εσμπολά από το Ιράν και ότι ε, το επέτρεπε αυτό ο Ασάντ. Όμως, εντωμεταξύ, τα πράγματα έχουν ησυχάσει στα σύνορα. Βεβαίως καλείστε να δραστηριοποιηθείτε σε άλλα επίπεδα. Έγινε τέτοιο ερώτημα της Τουρκίας. Διαπιστώνουμε από τη μια τους Πεσμέργα, τους Κούρδους Πεσμέργα στη Συρία που είναι οι καλύτεροι μαχητές ε, κατά του ISIS. Αυτούς όμως ε, τους μάχεται και τους αντιμάχεται η Τουρκία. Από την άλλη βλέπουμε να διαμορφώνεται μια κατάσταση Κατάσταση λοιπόν όπου το καθεστώς προσπαθεί με τη βοήθεια της Ρωσίας να στριμώξει τη μετριοπαθή αντιπολίτευση και κυρίως αυτούς ε, που βρίσκονται ε, στα σύνορα με την Τουρκία. Ε, ποια είναι η δική σας στάση, η μετριοπαθή της αντιπολίτευσης που έρχονται σε εσά τους σώζετε για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα από το καθεστώς ή όχι. Ας πούμε, επιτρέπεται τη διέλευση των συνόρων στους ασθενείς, γιατί ξέρετε με ενδιαφέρει να ξέρω ε, τι ακριβώς κάνετε σε σχέση με ανθρωπιστικής φύσεως προβλήματα. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τις σχέσεις με το Ιράν, ε, το να υπάρχει μια συμφωνία με το Ιράν ή όχι, εκεί δίστανται οι απόψεις. Νομίζω ότι η περισσοτερη Ισραηλινοί πολιτικη είναι κατά αυτής της συμφωνίας. Εγώ, αλλά και οι περισσότεροι εδώ στο Κοινοβούλιο, τίνουμε να πιστεύουμε ότι είναι καλό που υπάρχει αυτή η συμφωνία και εντωμεταξύ διαπιστώνουμε ότι το Ιράν ε, επιθυμεί κάποιες ε, σχέσεις ε, σε επίπεδο τεχνολογικό. Δεν πιστεύετε ότι αυτό το βήμα που έγινε ανοίγει μια προοπτική έτσι ώστε και εσείς στο μέλλον να μπορείτε να αναπτύξετε με το Ιράν άλλου είδους σχέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εσείς ε, ηγείστε μιας ε, πολύ ενδιαφέρουσας επιτροπής στο Κοινοβούλιο. Ε, ασχολείστε με θέματα άμυνας και ασφάλειας και έχω να υποβάλω τρεις ερωτήσεις. Και εδώ θα ήθελα να συνεχίσω ε, από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Γκάλα. Αντιμετωπίζει διάφορες απειλές, μεταξύ αυτών το Ιράν. Όσον αφορά τα... τον απλισμό στο Ιράν ε, μεγάλου βεληνικούς Θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι πρέπει να καταστραφούν αυτά τα όπλα, γιατί υπάρχουν δύο λύσεις. Εσείς ε, πώς αξιολογείτε την απειλή από το Ιράν όσον αφορά στα πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι τι ε, γίνεται με το θέμα της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων. Το άλλο θέμα είναι η Συρία. Κοιτάξτε, η ιστορία δείχνει ότι το, το Γκολάν εκεί έχουν ε, ε λάβει χώρα πολλές πολεμικές αντιπαραθέσεις. Ποια είναι τώρα η κατάσταση στα ψώματα του Γκολάν. Στη Συρία Έχουμε ε, διάφορες καταστάσεις ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται κανεί. Και η τρίτη ερώτηση είναι η εξή. Αυτό είναι κάτι που με απασχολεί πραγματικά. Δηλαδή έχουμε την δύναμη του Ισραήλ που απορρέει όχι μόνο από το γεγονός ότι είσαστε μια χώρα που έχει ε, πάρα πολύ καλά οργανωμένο το σύστημα ε, των μυστικών υπηρεσιών αλλά έχετε και τεχνολογική υπεροχή. Ε, μπορείτε να διεξάγεται πολέμους ε, με χειρουργική ακρίβεια. Ε, νομίζω οι λύσεις που προτείνετε εσείς εξακολουθούν να είναι καλύτερες στον κόσμο. Πάντως ε, υπάρχει, μένεται πόλεμο στη γειτονιά σας, στη Συρία και αυτό δείχνει επίσης και τα αποτελέσματα της τεχνολογίας. Αν δούμε λοιπόν το όλο θέμα κάτω από τεχνολογικό πρίσμα, ας δούμε λιγάκι την αεροπορία. Έχουμε διαφορετική τεχνολογία στην Αμερική, διαφορετική στη Ρωσία, στην ρωσική αεροπορία, το θέατρο του πολέμου. Εκεί δοκιμάζονται οι τεχνολογίες. Βλέπετε να διαφαίνονται νέες λύσεις. Γιατί κάθε πόλεμος δείχνει κάτι. Και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να φανούν οι τεχνολογίες που έχουν απτυχθεί για πολεμικές αντιπαραθέσεις. Κύριος Φρουντζούλητσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι η σταθερότητα και η ειρήνη ποτέ δεν δεχόταν τόσες απειλές όσο σήμερα. Μιλώ βέβαια για την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντιμετωπίζουμε τόσες απειλές και τόσες προκλήσεις ε, στον τομέα της ε, άμυνας ε, και της ασφάλειας και αιτίως να λάβουμε υπόψη ότι μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική σχέση. Έχουμε κοινά συμφέροντα για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Πώς βλέπετε, με επιθυμή παρέμβαση ε, Τουρκία, της Τουρκίας και της Αραβίας με στρατεύματα στη Συρία. Πώς θα επηρεάσει αυτή την κατάσταση, ιδίως μετά τη ρωσική επέμβαση που περιέπλεξε κατά πολύ την κατάσταση. Δεύτερον, το Ισραήλ και επαγγελματίες, α το πω έτσι, πώς βλέπουν αυτό το τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ευρώπη. Πώς θα επηρεάσει αυτό την σταθερότητα και την ειρήνη, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, φαίνεται ότι το ίσις έχει στην κατοχή του χημικά όπλα. Πώς θα συγκρατήσει την τεράστια αυτή απειλή για την ασφάλεια και για τη σταθερότητα του Ισραήλ. Ευχαριστώ κύρια Βάκμανς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ κάθομαι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας ε, σήμερα το μεσημέρι. Οι ερωτήσεις μου είναι παρόμοιες με αυτές των συναδέλφων που προηγήθηκαν στο λόγο. Πρώτα η κατάσταση στη Συρία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω την εμπλοκή της Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας ε, στη Συρία πώς τη βλέπετε. Και όπως και άλλοι συνάδελφοι, και εγώ ρωτώ πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το ίσις. Είναι σημαντικό το θέμα, θέλω τη γνώμη σας. Τρίτον, ε, βέβαια, η κρίση του μεταναστευτικού για εσά ποιε είναι οι βασικέ επιπτώσει ε, τη μεταναστευτική κρίση για τη χώρα σα και για τη Μέση Ανατολή εν γέννη. Θα θέλαμε να ακούσουμε τι απόψει από αυτό. Ευχαριστώ. Η ε, Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις έχουν ήδη ερωτηθεί, άρα είναι δύσκολο να θέσω και εγώ τώρα κάποιο ερώτημα. Αν μου επιτρέπετε να καλωσορίζω για μια ακόμη φορά ε, θέρμα τον πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να καλωσορίσω και όλους τους ε, βουλευτές της ΚΝΕΣΕΤ. Έχω πάντως ε, να κάνω κάποια ερωτήματα κι εγώ. Πώς περιγράφεται την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία. Ένα άλλο ερώτημα είναι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ με αυτά τα μαχαιρώματα είναι κάτι καινούριο. Δεν το είχαμε ξανακούσει, δεν ξέρω, μπορεί για εσάς να μην είναι κάτι καινούριο, θάνατοι από μαχαίρωμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση ο Πούτιν παρουσίασε πρόσφατα ε, την πρόταση για έναν ε, συνασπισμό στη Συρία με ε, την παροχή πληροφοριών ως πρόσφορα και ανέφερε και τρεις άλλες χώρες, Ιράν, Ιράκ, είπε η πρόεδρος, ως, πρόεδρο, ως πηγές πληροφοριών. Ίσως υπάρχουν ιρανικές απώλειες ε, στη Συρία. Μπορεί να έχουμε κάποιο πρόβλημα με την ενημέρωση. Εσείς ε, τι σενάρια εξετάζετε ε, για τη Συρία αρκούν οι αεροπιδρομές, μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και χερσαία παρέμβαση από ειδικές δυνάμεις ίσως. Υπάρχει όμως και μία ακόμη ε, συνάδελφος θα ήθελα να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, κυρία Άννα Γκόμες. Εκτός μικροφώνου, κυρία Γκόμες. Welcome. Ε, ε, ε. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε και να καλωσορίσω και τα άλλα μέλη της Κνεσέτ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Με αυτά τα μαχαιρώματα αλλά ε, υπάρχει και κάτι που ανησυχεί εμένα ακόμη περισσότερο για το μέλλον και για την επιβίωση, αν θέλετε, του Ισραήλ. Είναι το γεγονός ότι όλο και περισσότερο μορφωμένοι νέοι από την Παλαιστίνη είναι τόσο απεγνωσμένοι, απελπισμένοι, που λένε δεν θέλουμε μία λύση με δύο κράτη, αλλά ένα κράτος μόνο. Δίνουμε όλα τα δικαιώματα στο Ισραήλ. Αλλά αυτοί που δεν μαχαιρώνουν αλλά σας λένε ότι αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί έτσι, ε, είναι μια ελκυστική ιδέα αυτή. Τι είναι η άποψη, ποια είναι η άποψή σας. Επίσης θα ήθελα ε, και εγώ να ακούσω ε, τις απαντήσεις ε, στα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα που σας υποβλήθηκαν για το πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση στη Συρία. Εσείς στη Συρία πού είστε. Βλέπετε τι γίνεται, το χάος που κρατεί γύρω σας και λέτε καλύτερα να είμαστε εμείς έξω από το μάτι του κυκλώνα ή έχετε κάποιο άλλο ρόλο. Ποιος είναι ο ρόλος σας. Ανούς Ραγκά ήταν στο, σε κάποιο νοσοκομείο στο Ισραήλ. Υπήρξε κάποια άλλη είδηση ότι εργάζεστε ε, ε, για τον Άσαντ μαζί με την ε, Ρωσία. Μετά ακούσαμε για το Ιράν που δεν είναι και φίλος της Τέλο πάντων. Ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Ζαρίφ, χθε στο Κοινοβούλιο και μας είπε γενικώ ότι ε, είναι εκρηκτική κατάσταση. Και σε άλλους τομείς δεν υπάρχει μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπάρχουν και άλλα προγράμματα πυρηνικά και μη που δεν τα ελέγχει κανείς και θα μπορούσαν να ε, προκαλέσουν ε, καταστροφές απερίγραπτες στην ευρύτερη περιοχή. Και θα ήθελα τέλος να σας αναφέρω ότι σήμερα το πρωί παρακολούθησα ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα για ένα φάρμακο, ένα αρκωτικό που χρησιμοποιούν όλοι οι τρομοκράτες ε, μαχητές και φαίνεται ότι έχει ένα τρομερό ε, ε, αντίπτυχο, στη νεολαία. ναι, είναι έδωσαν φεταμίνης, πλέγεται κάπταγκον ή κάπως έτσι. Δεν μιλάω για την νεολαία, τον, ε, τους Ισραηλινούς νέους, γενικώ τους νέους μιλάω. Δεν θα οδηγήσει μεγαλύτερη αποξένωση και ριζοσπαστικοποίηση ο πρόεδρο. Πρέπει μάλλον το δοκιμάσουμε αυτό το νοικοτικό. Ήμασταν νέοι και εμείς κάποτε. Ναι, θύζει, είναι θυστικό όμως, ξέρετε, λέει η κυρία Η πρόεδρος. Υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει το λόγο, ναι. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να επωφεληθώ από την παρουσία σας εδώ για να μάθω περισσότερα πράγματα. Τα περισσότερα βέβαια ρωτήθηκαν από τους προλαλήσαντες. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε το εξής εμείς. Βλέπουμε να ε, ήταν στο σημείο μουσουλμανική αδελφότητα, τώρα είναι το ίσις στην εξουσία εκεί η σταθερότητα της πολιτικής κατάστασης στην Αίγυπτο ε, πώς έχει, πώς την αντιλαμβάνεστε. μετά την αλλαγή της κατάστασης ε, και μετά την ανατροπή του Μόρση, τι, τι έχει γίνει. Πώς έχει κατάσταση στη χώρα πολιτική. Γιατί ήταν πολύ μικρή η της κυβέρνησης αυτής και Τώρα να πω κάτι άλλο. Είμαστε διαρρεμένοι στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το ψήφισμα για την Παλαιστίνη το περσινό. Αυτό το ψήφισμα ή άλλα κείμενα του Κοινοβουλίου πώς έχουν επηρεάσει τις εσωτερικές συζητήσεις και πώς έχουν επηρεάσει και τις προοπτικές των ειρηνευτικών ε, συνομιλιών και διαπραγματεύσεων. Η διαδικασία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής αυτονομίας. Τώρα, αυτές οι επιθέσεις με τα μαχαίρια ε, τι δυναμική έχουν και επίσης και το θέμα της μετανάστευσης είναι ενδιαφέρον αλλά αναφέρθηκα από άλλους Πρόεδρος Εδώ θα κλείσω τον κατάλογο ε, των ομιλητών για να ε, μπορούν να ελέγχουν κάπως το χρόνο. Έχετε εσείς κύριε Πρόεδρε της Κνεσέτ. Τι ώρα πρέπει να τελειώσουμε. Okay. I brought sleeping bag. Έχω φέρει και το sleeping bag μαζί μου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ, θα κοιμηθώ εδώ. Γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Be, uh, as, as θα προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος και να εστιαστώ στις ερωτήσεις. Είναι πολλές ερωτήσεις ε, οι οποίες αφορούν τη Συρία, οι οποίες αφορούν την Τουρκία, άλλες για την, ε, το Ιράν, την Αίγυπτο. Θα τα δούμε. Είναι, είναι τα διάφορα στοιχεία τα οποία αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Να ξεκινήσουμε από τα καλά. τα καλά κατά τη δικιά μας άποψη είναι η Αίγυπτος. Όταν ε, η μουσουλμανική αδελφότητα ε, ανέλαβε τα ενία της Αιγύπτου δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αλλά αρκετά σύντομα, αρκετά γρήγορα διαπιστώσαμε, συνειδητοποιήσαμε ότι αναμφίβολα η Αίγυπτος θέλει ε, ήθελε να ε, λήξει η συμφωνία του 78 ανάμεσα ε, στην Αίγυπτο και το ε, Ισραήλ. Γιατί στους πολέμους του 56, του 67, του 73 έχει ε, ε, ε, πολλές εκατοντάδες Ισραηλινοί και Αιγύπτιοι έχασαν τη ζωή τους και τότε ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ και ο πρόεδρος Αιγύπτου Σαντάτ μας έσωσαν με αυτήν την συμφωνία η οποία λειτουργήσε για 40 χρόνια σχεδόν και ξαφνικά, ξαφνικά ε, άρχισε να δυναμητίζεται και σκεφτήκαμε ότι θα ξαναρχίζαμε πάλι την ίδια κατάσταση όπου θα έπρεπε ένα τρίτο του προϋπολογισμού μας να αφορά τα στρατιωτικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Αίγυπτο, ε, να έχουμε ε, χιλιάδες τάγκς στο Σινά όπως γινόταν παλιά και αυτό ήταν πάρα πολύ αξιογόνο για μας αλλά τα πράγματα άλλαξαν ε. και ξαφνικά είχαμε μία ε, ευτυχή έτσι, εξέλιξη της ε, αναταραχής και ένας θαραλέος ηγέτης, ο Αλφατ Ασίση, ανέλαβε τα ημεία και εκπροσώπησε όλα αυτά τα λογικά έθνη που θέλουμε να δούμε την ε, ψύχρεμη διπλωματία να αναλαμβάνει. Και ε, λόγω και της ε, ανάπτυξης του ISIS είδαμε έτσι μια καλή εξέλιξη όσον αφορά την ασφάλεια σε σχέση με την Αίγυπτο γιατί και εκείνοι απειλούνται όπως και εμείς από το Ισλαμικό κράτος. Και μετά από 70 χρόνια ειρήνης θεω θεωρήσαμε ότι ήταν ε, μια ψυχρή ας πούμε ειρήνη. Ε, ε, φαινόταν να συνειδητοποιούν ότι το Ισραήλ είναι τέρος και εμείς ξαναανακτήσαμε την κυριαρχία στο Σινά. Δηλαδή εννοώ την, εννοώ ότι κατάλαβαν ότι δεν μας χρειάζονται. Βεβαίως αν μας χρειαστούν εντάξει θα ε, ε, βοηθήσουμε, αλλά ε, πληρώνουν βαρύ τίμημα για το, στον ISIS και στο Κάιρο και αλλού έχουν κάθε μέρα θύματα. Πρόκειται για ένα θέμα που είναι σημαντικό και για αυτού και για μας και του ευχόμαστε τα καλύτερα έτσι ώστε να μπορέσουν να πολεμήσουν κατά του ISIS γιατί πραγματικά πολεμούν ε, με έναν πραγματικό φυσικό εχθρό κάθε μέρα. Αυτό είναι τα καλά νέα. Όλα τα άλλα όπως γνωρίζετε είναι η μία τραγωδία μετά την άλλη. Στην Ιεμένη, στη Λιβύη, στο Ιράν και ίσως ε, σκληρότερα ακόμα στη Συρία. 470.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ε, ε, πολλοί μεταξύ αυτών είναι παιδιά. Δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Έχουν γίνει πρόσφυγες. Άλλοι, έχουν εκτοπιστεί εντός της Συρίας. Ζουν ακόμα στη Συρία, αλλά η Συρία δεν είναι πια όπως ήταν. Έχουμε πολιτοφυλακές ε, που ε, δρούν σε ολόκληρη την επικράτεια και αν με ρωτάτε δεν νομίζω ότι είναι κανείς προφήτης να μπορεί να ξέρει τι θα γίνει και πώς θα, είναι, πώς θα λήξει αυτή η κατάσταση. Ωστόσο, είναι κάτι που θίγει την Ευρώπη και την, αφορά και την Ρωσία ε, και βεβαίως είναι σημαντικό το θέμα και για το Ισραήλ. Αναφέρθηκε και εδώ προηγουμένως ε, ότι εμείς ε, στην ουσία βρισκόμαστε ε, από το 1972 και μετά δεν είχαμε συμβάντα ας πούμε περίεργα στα σύνορά μας με την γειτονική χώρα και τώρα βλέπουμε έχουμε πολλά προβλήματα ε, βλέπουμε να περνάνε πύραυλοι, βλέπουμε να περνάνε οπλικά συστήματα, να πηγαίνουν προς τη Συρία ή από το Συρία στο, ε, στο Λίβανο. Ε, οπωσδήποτε υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να μας επιβληθεί για μία ακόμα φορά ο διαρκής πόλεμος. ωστόσο παρόλα αυτά ήταν τα, τα σύνορα ήσυχα Τώρα όμως ε, τα πράγματα άλλαξαν. Στον Κόλεχαν έχουν χάσει τον έλεγχο ε, των συνόρων ε, και έχουμε τις ομάδες των τρομοκρατών οι οποίοι προσπαθούν να προχωρήσουν το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μία buffer zone ανάμεσα από το χάος και την χώρα μας. Ένα, ε, ε, ε, μία δηλαδή περιοχή ανάσχεσης Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως και εμείς ξέρετε ότι οι στρατιώτες μας ήταν όλοι πολίτες πριν γίνουν ε, στρατιώτες λόγω της ε, κατάστασης και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε ε, τα πράγματα γιατί είναι τόσες πολλές παραστατικές οργανώσεις που δεν ξέρουμε ακριβώς, πρέπει να τις πολεμήσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε όλες. Οπωσδήποτε ε, μέχρι τώρα ε, έχουμε σώσει πολλές ζωές γιατί ε, είχαμε στα σύνορα μια καλή οργάνωση και χαιρόμαστε γιατί καταφέραμε να βοηθήσουμε. Έχουμε ανθρώπους που περνούν τα σύνορα διαρκώς. Είναι σημάδι του πολέμου που συνεχίζει και συνεχίζει. Έχουμε τώρα δύο απειλές από το Ισλαμικό κράτος ε, ε, στο Σινά, η Άνσερ Μπέτελ και έχουμε και το και μάλιστα έχουν δεσμευτεί να, στο πλευρό του Ισλαμικού κράτους ε, χρηματοδοτούνται από το Ισλαμικό κράτος τους ε, ε, αντιμετωπίζουν κυρίως τον ε, Αιγυπτιακό στρατό, αλλά σίγουρα όταν αισθανθούν ότι έφτασε η ώρα θα στραθούν και εναντίον μας. Από την πλευρά της Συρίας έχουμε μια άλλη ομάδα, είναι η Σουχαντάλη Αρμούκ, έχουν πάρει το όνομά τους από ένα ποτάμι που βρίσκεται ανάμεσα στο Ισραήλ, τη Συρία και το Λίβανο και αυτοί είναι ορκισμένοι ε, σύμμαχοι ε, του Ισλαμικού ε, κράτους, καταφέρονται κατά του Ασάντα και του καθεστώτος του. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι το Ισλαμικό κράτος δημιουργεί προβλήματα όχι μονάχα με τις επιθέσεις που κάνουν παντού, στο Βέλγιο, στο ε, τουλάχιστον μία φορά στην Γαλλία αλλά και αλλού. Ε, εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και σε άλλα ε, μέτωπα και επομένως μέσω κατασκοπίας, μέσω συλλογής πληροφοριών πρέπει να είμαστε σε θέση να τους αντιμετωπίσουμε και να τους περιορίσουμε. Εμείς ε, βλέπουμε ότι η γενική κατάσταση έχει αλλάξει μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας τα 40 τελευταία χρόνια. Αρχικά ε, το φιλοσοφικό μας, έτσι, το αμυντικό μας δόγμα ήταν ότι θα πρέπει να σώσουμε ε, την χώρα μέσω του στρατού, να μην χάσουμε κανένα πόλεμο, γιατί εμείς κάναμε δεκάδες πολέμους, αλλά θεωρούσαμε ότι αν χάσουμε έναν θα ήταν το τέλος του κράτους του Ισραήλ δηλαδή ε, συμβατική μάχη κατά των στρατών. Ε, γιατί οι απειλές ήταν πολλές για το νεαρό και νέο συσταθέν κράτος του Ισραήλ από το 56, μετά το 67, μετά το 73. Μετά όμως η κατάσταση άλλαξε. Ε, δεν είχαμε ε, πλέον ανάγκη για πολέμους με συμβατικό στρατό. Είχαμε δύο ε, συμφωνίες ειρήνευσης οι οποίες, ε, οποίες λειτουργούσαν με την Αίγυπτο και με την Ιορδανία. Τώρα όμως μας περικυκλώνουν πέντε τρομοκρατικές ομάδες, η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντα στην Γάζα. Έχουμε τον Ισλαμικό στρατό και στα υψώματα του Γκολάν και στην Αίγυπτο, η Αλκάιντα και η Χιντάλα στο βορρά έξι επομένως είναι η not an uh, Και η Χεσμολά. Ε, ε, έξι λοιπόν είναι οι τρομοκρατικές ε, ε, οργανώσεις ε, οι οποίες αποτελούν ασύμετρες ε, απειλές για μας και δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ποια είναι τα, ποιοι είναι οι περιορισμοί που τίθενται από ένα πόλεμο τέτοιου είδους. Έχουμε τώρα και άλλους πολέμους, έχουμε εχθρούς διαφορετικούς, από το facebook. Μην γελάτε γιατί πραγματικά, ξέρετε, ξυπνάει κάποιος, γράφει κάτι στο facebook που λέει ας πούμε ότι σήμερα ε, θα ε, γίνουν μάρτυρες κάποιοι γιατί πριν από τρεις μέρες ένας Ισραηλινός στρατιώτης προσέβαλε ε, έναν ξάδερφο τέλος πάντων και έχασε κάποιος τη ζωή του και θέλουν να γίνουν μάρτυρες. Δεν ανήκουν σε καμία ομάδα, ε, είναι μοναχικοί, είναι μεμονωμένοι, δεν τους πιάνουν ε, οι υπηρεσίες ας πούμε ε, πληροφοριών, δεν υπακούν σε κάποιον αρχηγό που έχει την έδρα του στη Συρία αλλού, πηγαίνει στην κουζίνα της μάνας του, παίρνει ένα μεγάλο μαχαίρι και το χρησιμοποιεί έτσι ώστε να προσπαθήσει να ε, τραυματίσει άμαχους ε, είτε οποιονδήποτε άλλον. Απλώς δηλαδή προσπαθεί να κάνει κάποιο θύμα, να προκαλέσει ε, ε τέτοιου είδους δράση, γιατί αισθάνεται ότι γίνεται μάρτυρας εάν σκοτωθεί στη διάρκεια μιας τέτοιας προσπάθειας, ενός τέτοιου συμβάντος. και ε, από τη μία πλευρά βεβαίως ε, οφείται από την ε, απελπισία γιατί βλέπω ότι δεν αλλάζει η κατάσταση, από την άλλη κάποιοι τον βάζουν να κάνει, τον ενθαρρύνουν να κάνει κάτι τέτοιο με εργαλεία όπως είναι το facebook, όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα που με, με τα γλαφυρότερα χρώματα παρουσιάζουν τέτοιου είδους κινήσεις. Είχαμε πάρα πολλά μαχαιρώματα, ας πούμε, τους τελευταίους μήνες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, παρόλα αυτά την αντιμετωπίζουμε. Είμαστε μια ισχυρή ε, κοινωνία. Ξέρετε ότι εμείς γίναμε ένα εργαστήριο εκμάθησης της ε, της αντιμετώπισης του τρόμου ε, και έχουμε μάθει πώς να τον αντιμετωπίζουμε τον τρόμο αυτό. Πριν από 10 χρόνια είχαμε τους καμικάζι, οι οποίοι επιτίθενται όχι με μαχαίρια, αλλά με αυτοσχέδιες βόμβες ε, και περίπου 500 άνθρωποι ε, έχασαν τη ζωή τους πριν από δύο περίπου χρόνια. Πάει αυτό, τελείωσε βέβαια, γιατί τώρα ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο των ε, βομβιστών αυτοκτονίας. Ξέρουμε πώς να τους εξουδετερώσουμε. Και παλαιότερα είχαμε και το πρόβλημα ε, των Ισραηλινών που ε, πήγαν στο εξωτερικό το 1972 ας πούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου αργότερα με απαγωγές, με αεροπειρατείες το θέμα βέβαια δεν είναι για μας ε, να αντιμετωπίζουμε εκ των υστέρων την τρομοκρατία αλλά εκ των προτέρων να σταματήσει ο πόλεμος με την Παλαιστίνη αυτή η διαμάχη που διαρκεί χρόνια. Και έτσι λοιπόν φτάνω στην ουσία του προβλήματος την ευρωπαϊκή συμβολή ή μη συμβολή στα τεκτενόμενα. Εμείς πιστεύουμε ότι η συμφωνία που συνάψαμε με την Αίγυπτο και με την Ιορδανία ε, με αυτήν μπορούμε να συνάψουμε συμφωνία και με τους ε, Παλαιστίνιους. Ήδη άνθρωποι είναι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που και αυτοί έχουν την ε, προσδοκία της ζωής, έχουν συναισθήματα. Αλλά σας λέω, για να γίνουν όλα αυτά ε, πρέπει να υπάρχουν ηγετικές φυσιογνωμίες. Ας πούμε, ο βασιλιάς Χουσέιν ήρθε στην Ιερουσαλήμ και έκατσε τότε παλαιότερα με τον Πρωθυπουργό Ραμπίν και υπέγραψε μια συμφωνία που ήταν επωφελής και για τις δύο πλευρές. Μετά ο Σαντάτ είχε το τάρος να έρθει στην Κνεσέτ, να απευθυνθεί στους Ιζαλινούς, να τους κερδίσει, να μιλήσει στην καρδιά τους, να τους εξηγήσει ότι δεν θα παρετηθεί από τις διεκδικήσεις του ήταν ρεαλιστής και για το ΣΥΝΑ δεν έλεγε ότι θα πετάξει, διώξει όλους τους ε, Ισραηλινούς από το ΣΥΝΑ, ούτε έλεγε ότι το ΣΥΝΑ θα ε, προσαρτιστεί, θα ενταχθεί στην Αίγυπτο. Έλεγε και είπε όμως να μην χυθεί άλλο αίμα. Και έτσι λοιπόν ενέπνευσε και σε εμάς την αίσθηση του συμβασμού. Να πούμε ότι ε, κάνουμε παραχωρήσεις για κάποιον με σωστό όραμα για το λαό του. Τώρα, με τους Παλαιστίνιους για πάρα πολλά χρόνια είμαστε άτυχοι. Δεν έχουμε τέτοια ηγετική φυσιογνωμία. Όπως ξέρετε, ο Αραφάτ ε, για πάρα πολλά χρόνια ήταν μέσα σε δύο βάρκες. Προσπαθούσε να μιλάει πολιτισμένα θα το χαρακτηρίσω, αλλά κατ' ουσίαν την τρομοκρατία. Πάει ο Ρασάτ, ο Αμπού Μαζέν Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσά τον έχετε συναντήσει. Εγώ τον έχω συναντήσει δύο φορές. Πιστεύω ότι είναι κάποιος που λέει αυτό που πιστεύει είναι κατά της βίας, σαφώς κατά της ε, τρομοκρατίας και κατά κάποιο τρόπο αυτή είναι η ηγετική φυσιογνωμία που χρειαζόμαστε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν έχει τη δύναμη που θα έπρεπε να έχει γιατί τους μισούς Παλαιστίνες δεν του ελέγχει οι μισοί είναι στη Γάζα και αυτούς ελέγχει η Χαμάς. Και αυτοί είναι κατά όλων αυτών που πιστεύουμε και εμείς και όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ, κατά της ειρήνης, ε, υπέρ της βίας, υπέρ της τρομοκρατίας. Αυτοί δεν θέλουν συμβασμό γιατί πιστεύουν ότι το δικό τους το όρομα είναι να μην πάψουν να αγωνίζονται μέχρι να εξαλωθούν, να εξαφανιστούν οι, άπι, άπιστοι. Ο Αμπού Μαζέν τους μισούς όπως σας είπα δεν τους ελέγχει και τους άλλους μισούς που είναι πιο ρεαλιστές εκεί δεν προχωράει όσο πρέπει να κάνει μεγάλη παραχώρηση έτσι ώστε να κάνει αυτό που κάναμε εμείς. Δύο από εμά είναι στην αντιπολίτευση, δύο είναι πιο αριστερά. Αλλά ακόμα και η αριστερά στο Ισραήλ δεν μπορεί να δεχτεί αυτό που ορίζουν οι Παλαιστίνοι ως το δικαίωμά τους της επιστροφής, δηλαδή να κατακλείσουν το Ισραήλ με πρόσφυγες που έφυγαν από το 48 ακόμα και τους πρόγονους τους. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα ότι ο Παλαιστίνιος ηγέτης πρέπει να πει στο λαό του, κοιτάξτε, τώρα τέλειωσε αυτό το όνειρο, δηλαδή η Παλαιστίνα κατακλείσει όλη αυτή την περιοχή και το μικρό Ισραήλ. Θα λύσουμε το πρόβλημα των Παλαιστίνων προσφύγων στην Παλαιστίνη και όχι στο Ισραήλ. Για να γίνει αυτό θα έπρεπε να λάβει χώρα μια πραγματική μεταμόρφωση σε μια ηγετική φυσιογνωμία Παλαιστινίου και κάτι τέτοιο θα οδηγούσε, αν όχι αμελητή, σίγουρα σιγά σιγά σε κάποιες ε, διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να αποκληθούν ιστορικός συμβασμός. Το Ισραήλ και με δεξιά ηγεσία έχει δεχτεί αυτή τη λύση των δύο κρατών. Ο Πρωθυπουργός ίσως κανείς να μην τον πίστευε, αλλά ήδη το 2009 που τότε ήταν ε, υπουργό, ε, μίλησε για τα δύο κράτη και σας διαβεβαίω δεν θεωρεί ότι υπάρχει λύση. Είπε κάποια κυρία ότι ε, ποια είναι η λύση. Μα αν υπάρχει μόνο ένα κράτος, αυτό σημαίνει ότι εξαφανίζεται το κράτος του Ισραήλ. Η άλλη λύση είναι να συνεχίζεται στο διηνεκές ε, ο πόλεμος, να ε, σκοτώνουμε και να σκοτωνόμαστε και δεν μπορεί αυτό να είναι το όραμά μας. Σιγά σιγά ολοκληρώνω, πολύ ευχαρίστω. Έτσι λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι αυτά πρέπει να γίνουν. Ο ρόλος της Ευρώπης, πρέπει να είμαι μαζί σας, ο ρόλος της Ευρώπης πρέπει να είναι όχι να αποθαρρύνει τους Παλαιστίνιους για να απεμπολίσουν την ιδέα των άμεσων διαπραγματεύσεων. Του αντίον να τους ενθαρρύνει να επανέλθουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Γιατί αν τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν και νομιμοποιούν το Παλαιστινιακό κράτος χωρίς όμως οι Παλαιστίνοι να συμβαστούν μαζί μας και αν τους ε, λένε ότι ξέρετε μπορείτε να πάτε στο ε, Συμβούλιο Ασφαλείας ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, τους τα λένε αυτά και ξέρετε γίνεται παρακάμπτονται οι διαπραγματεύσεις και ο διάλογος, ο οποίος όμως είναι εκείνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τέλος της σύγκρουσης. Αν λοιπόν η Ευρώπη θέλει να εμπλακεί, πράγμα που εγώ επιθυμώ διακαώς, η Ευρώπη μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα, να φτιάξει τις γέφυρες, αλλά πρέπει να πείσει τους Παλαιστίνιους ότι κανείς δεν μπορεί να τους δώσει κράτος χωρίς να υπάρχει το Ισραήλ. Το Ισραήλ πρέπει να συμμετέχει διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν από μηδενική βάση και μετά μπορούν οι Ευρώπαιοι να διαμεσολαβήσουν, όλοι μπορούν να μας βοηθήσουν, αλλά όχι με έναν τρόπο που θα είναι αντιπαραγωγικός. Κάθε άλλο πρέπει να καταλάβουν ότι οι Παλαιστίνοι πρέπει να επανέλθουν στην τράπεζα των υπραγματεύσεων. Το τέλος, τελευταία παρατήρησή μου για το Ιράν. Δεν χρειάζεται να σε εξηγήσω γιατί αποτύχαμε. Ε, τέλος πάντων, αυτά όλα ανήκουν στο παρελθόν. Αυτό όμω που δεν ανήκει στο παρελθόν είναι ότι η συμφωνία που υπογράφηκε πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση για να είμαστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζεται. Η Ιρανοί είναι, έχουν πείρα το να χαράζουν μια κόκκινη γραμμή, μετά να την κομματιάζουν σε ροζ γραμμούλες και να παραβιάζουν κατά καιρού αυτές τις ροζ γραμμούλες, όπου δεν προκαλούν κανένα, αλλά κάποια στιγμή όλοι διαπιστώνουν, μα δεν υπάρχει πια κόκκινη γραμμή, την έχουν παραβιάσει οι Ιρανοί. Το έκαναν όμω με πολύ ήπιο και υφέρποντα τρόπο. Ας είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν δική μας χαρά να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστούμε πολύ την αντιπροσωπεία που μας επισκέφτηκε. Θα περάσουμε εντός ολίγου στο επόμενο θέμα της διάταξης.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 Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την αυτοεξοχότητα τον πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Κέιτσι Κατακάμι. Να καλωσορίσω επίσης τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της Ιαπωνίας, τον κύριο Σίγκο Γιαμαγκάμι σημερινό θέμα, στην ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε, είναι η νέα νομοθεσία της Ιαπωνίας για την ασφάλεια και την ειρήνη. Το Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς υιοθετήθηκε και για μας συνιστά μια μείζων αλλαγή Το αμυντικό δόγμα ε, και στην πολιτική εξωτερικών της Ιαπωνίας. Θα μας ενδιαφέρει λοιπόν να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και να συζητήσουμε το ζήτημα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Έχει πέρασει αρκετό καιρό την τελευταία φορά που το συζητήσαμε το θέμα, γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα με την παρουσία των δύο αξιότιμων προσκεκλημένων μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you ευχαριστώ πολύ και να καλησπερίσω τους παρισταμένους. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την ε, Φωτίγκα, κυρία Φωτίγκα, την πρώτη επιτροπή και τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους της που με καλέσετε να μιλήσω για τις σχέσεις ε, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εστιάσω βέβαια στα θέματα της ασφάλειας και θα δώσω στη συνέχεια το λόγο στον κύριο Γιαμαγκάμι. Σήμερα θέλω να σας πω ότι οι σχέσεις Ιαπωνίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Σήμερα έχουμε στενές σχέσεις ε, που βασίζονται σε μια ισχυρή δέσμευση ε, στις αξίες της κόνης αγοράς, της δημοκρατία, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας. Ε, σήμερα συνεργάζονται η Ιαπωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλούς τομείς που υπερβαίνουν κατά πολύ τους παραδοσιακά ισχυρού δεσμού που είχαμε ανέκαθα στον τομέα των εμπορίων και των επενδύσεων. Ένα από του βασικού τομεί όπου η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών έχει αναπτυχθεί τα μάλλα είναι ο τομέα ε, της ειρήνης και τη ασφάλεια. Βασιζόμαστε σε κοινέ αρχέ και σε κοινέ αξίε. Ε, και έτσι έχουμε σφυριλατήσει μια ισχυρή σχέση στον τομέα αυτό και συνεργαζόμαστε στενά για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στη διεθνή κοινότητα. Η ανάπτυξη των σχέσεων στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας ε, μπορεί να την αντιληφθείτε βλέποντας ε, τη συνεργασία ε, της Ιαπωνίας στην κοινή εξωτερική πολιτική πολιτική άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 14 για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Δύναμη ε, συνεργάζεται με την Αταλάντη, την ε, επιχείρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταβλέψη της ε, πειρατείας, για τον εντοπισμό πειρατών και έχουμε και κοινέ ναυτικές ασκήσεις στον κόλπο του Αντέν. Επίσης συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην, στο Μαλί, στον Ήγυρα και θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας στο κέρας της Αφρικής και στην Ουκρανία. Αυτά τα παραδείγματα νομίζω ότι είναι ε, προφανής ε, η συνολική αυτή η γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνάδει και με τη γενική στρατηγική της Ιαπωνίας για την ασφάλεια, δηλαδή μια ενεργητική συνεισφορά στην ειρήνη με βάση την αρχή της διεθνούς συνεργασίας. Πρόσφατα υπήρξε μια θετική εξέλιξη στο τομέα τη εργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία είπε και η πρόεδρο ότι το Σεπτέμβριο τη προηγούμενη χρονιά πέρασε από την ε, Ιαπωνική Βουλή ένα νέο νομοσχέδιο για την ασφάλεια και την ειρήνη. Ο συνάδελφος Γιαμαγκάμι θα επεκταθεί σε κάποιες άλλες ε, πτυχέ. Εγώ εδώ θα ήθελα να αναφέρω μόνο πώς η εν λόγω νομοθεσία θα δώσει στην Ιαπωνία τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε ένα ευρύ φάσμα ε, επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης, σε συντονισμένες διεθνείς προσπάθειες. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στην Ιαπωνία να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, να παρέχει υποστήριξη. Με αυτή την νομοθεσία νομίζω ο αντίκτυπος θα είναι ιδιαίτερα θετικός στη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνία στον τομέα της ασφάλειας. Νομίζω αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα από το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει η νομοθεσία μας ότι είναι ένας από τους βασικούς μας εταίρους στις διεθνείς τονισμένες μας προσπάθειες και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ε, με την ΕΠΑ ε, μια πολύ πιο στενή συνεργασία. Ποιο είναι το ιστορικό χρονοδιάγραμμα τώρα. Εκπονούμε τι λεπτομέρειε, συζητούμε τα διάφορα μέτρα και διαδικασίε που θα πρέπει να αναλυφθούν στο πλαίσιο αυτή τη νέα νομοθεσία. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, διότι πρέπει να λάβουμε πολύ προσεκτικά υπόψη ε, τι ανησυχίε που εκφράστηκαν και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κατανοήσουμε και την ε, άποψη τη κοινή γνώμη στην Ιαπωνία. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω τα σχόλια του Ναβάρχου της ΝΑΦΟ στην επιχείρηση Αταλάντη για την καταπολέμηση της ε, πειρατείας, ο οποίος είπε ότι παρότι γεωγραφικά απέχουν πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία, είμαστε παγκόσμιοι εταίροι σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχουμε κοινέ αξίες, δημοκρατία, έχουμε θαλάσσιο εμπόριο, έχουμε την ελευθερία της ναυσιπλοείας ως βασικές αρχές. Αυτή ήταν η ε, αναφορά του Ναυάρχου και υπόθηκαν αυτά τα λόγια μετά από την πολύ επιτυχημένη συνεργασία μας. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν που πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα και να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την διεθνή μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Ε, τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιαμαγκάμι για να μας κάνει τη δική του ε, παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλο προνόμιο που μπορώ να απευθύνομαι στην ε, υποεπιτροπή σας, ε, την υποεπιτροπή ασφάλειας και άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Ιαπωνίας και ε, μια ομάδα προβληματισμού για θέματα διεθνούς ασφάλειας και έχω έρθει εδώ για να σας δώσω διάφορες προσωπικές σκέψεις και απόψεις δρατώμενος αυτής της ευκαιρίας. Στην Ιαπωνία πολλοί αντιλαμβάνονται ότι η Ευρώπη ανησυχεί και ασχολείται κυρίως με θέματα που αφορούν το ανατολικό μέτωπο και το νότιο μέτωπο. Ως παγκόσμια δύναμη όμως δεν περιορίζεται σε αυτά τα μέτωπα, αλλά πρέπει να δει και άλλα. Ήθελα και εγώ λοιπόν να σας ε, μεταφέρω ως τροφή για συζήτηση τις δικές μου σκέψεις. Ε, σε δύο άξονες θα κινηθεί η ομιλία μου. Μην ανησυχείτε ότι θα σας αποκοιμήσω βέβαια, δεν θα μακρηγορήσω ιδιαίτερα. Ε, λοιπόν, το πρώτο, ο πρώτος άξονας είναι η περιφερική κατάσταση και το δεύτερο σκέλος είναι τι θα αλλάξει με τη νέα νομοθεσία της Ιαπωνίας για την ασφάλεια. Δεν προτίθεμαι βέβαια να αναφερθώ δεξιωτικά σε όλες τις διαφάνειες που είχα ετοιμάσει, αλλά θα εστιάσω σε ορισμένα ε, προεξέχοντα ε, σημεία. Πρώτα απ' όλα, στη σελίδα 1 την ε, Ανατολική Ασία. Έχουμε κάποιες ε, πολύ σημαντικές εξελίξεις. Και δεν μιλάω μόνο για την Ιαπωνία, αλλά και σε άλλες περιοχές, σε άλλα κράτη της Ανατολικής Ασίας. Τι εννοώ αυτό. Τι εννοώ ε, μάλλον με όλα αυτά. Στη δεύτερη διαφάνεια βλέπετε ένα χάρτη που μπορεί να είναι κάτι με τον οποίο δεν είστε εσείς εξοικειωμένοι στην Ευρώπη, αλλά οι Ιάπωνες είναι πολύ εξοικειωμένοι με αυτό τον χάρτη. Βρισκόμαστε σε μια αξιοζήλευτη θέση γεωγραφική, διότι τριγυριζόμαστε από τρεις ε, πυρηνικές δυνάμεις, Ρωσία, Κίνα, Βόρεια Κορέα. Αυτές οι χώρες όμως δεν έχουν μόνο πυρηνικά όπλα, αλλά και ένα μόνιμο στρατό που αριθμεί πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Επομένως, δεδομένων όλων αυτών των στοιχείων, ας δούμε τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Τέταρτη διαφάνεια. Κορεατική Χερσόνησος. Εδώ εξηγούμε την κατάσταση στην κορατική Χερσόνησο. Είναι ένα déjà vu ίσως για εσάς. Συνδυασμός πυρηνικών δοκιμών με τις λεγόμενες ε, εκτοξεύσεις ε, δορυφόρων. Και πάλι φέτος, ε, το Γενάρη και το Φεβράριο είχαμε τέτοιου είδους εκτοξεύσεις και πυρηνικές δοκιμές. Ποια είναι η διαφορά όμως ότι σήμερα Μιλάει για βόμβα υδρογόνου η Βόρεια Κορέα. Η σοβαρότητα όμως των συμβάντων αυτών δεν θα πρέπει ποτέ να υποτιμηθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα το βαθμό της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει πολύ και πολύ περισσότερο από άλλες χώρες μεταξύ των οποίων είναι το Ιράν. Αν τώρα στρέψουμε το βλέμμα μας ε, στην ε, θάλασσα της Νότιας Κίνας, στην έκτη διαφάνεια εδώ, βλέπετε κάποιες φωτογραφίες που ίσως για σας είναι γνωστές και δείχνουν την κατάσταση. και τη στρατιωτικοποίηση και τις διεκδικήσεις ε, τώρα στην 7. Εδώ βλέπετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον τρίγωνο που έχουμε χαράξει. Ο αντινάβαρχος συγκεκριμένα κόντα, φίλος μου, στην Ίσο Χάινα μπορούν ε, αεροπλανοφόρα να, ε, να ελιμενίζονται, αλλά δημιουργούνται τώρα και αεροδιάδρομοι σε κάποια νησιά στην Νότια Κίνα, στα άλφα της Νότιας στο Ρούτι, στο Φίρι Κρος Ρίφ και ίσως και στο Σκάρμπορο Σόλ στο μέλλον. Βλέπετε ότι εδώ μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ε, υδατικό ορίζοντα και τι γίνεται εκεί είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και τη Μαλαισία που είναι παράκτιες χώρες ε, και επηρεάζονται αλλά και οι γειτονικέ χώρες όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Ινδία. Και η Ευρώπη όμως θα επηρεαστούν διότι αυτή η θάλασσα της Νοτιάς Κίνας μας παρέχει σημαντικούς θαλάσσιους διάβλους επικοινωνίας. Αν θέλουμε να εξαγάγουμε ε, στη, αν θέλετε να εξαγάγετε μάλλον σε Ιαπωνία, Κίνα, στην Ανατολική Ασία, ε, Ινδονησία κτλ. Θα χρειαστεί να περάσετε από εκεί. Σίγουρα λοιπόν η ελευθερία της ναυσιπλοείας είναι κάτι που ενδιαφέρει τους πάντες. Γι' αυτό και χρειάζεται να δοθεί προσοχή από την Ευρώπη σε αυτήν την περιοχή. Επόμενη σελίδα, επόμενη διαφανή εδώ. Για να σας πω κάτι ε, Δεν σας λέμε ότι πρέπει να επιλέξετε μια από τις δύο πλευρές. Δηλαδή ε, η Ιαπωνία ή Κίνα ή η Κίνα. Όχι. Τι είδους διεθνούς τάξεως θέλουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλουμε να χαρακτηρίζεται από εκφοβισμό και από αλαζονία αυτή η διεθνή τάξη. Πρέπει να υπάρχει ισότιμη εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών αυτών. Καμιά χώρα δεν έχει το δικαίωμα τον ε, ομολογό να τον ε, χαρακτηρίζει με αυτόν τον τρόπο, με τέτοιου είδους διαφημίσεις. Όπως σε, ε, σε αυτή τη εφημερίδα από τις Φιλιππίνες που βλέπετε ότι εμείς φαίνεται να απεκονιζόμαστε ως κοντικιά και αστείοι. Ήταν μια διαφήμιση, παραλαμβάνω, σε μια εφημερίδα στις Φιλιππίνες. Και πραγματικά εμένα με εξέπληξε. Τώρα, πάλι ε, στην ε, θάλασσα στρέφομαι, στην, ανατολική, στην θάλασσα της Ανατολικής Κίνας. Βλέπουμε συνεχής ε, ε, παρίσφρηση ε, όλο και συχνότερη στα εδαφικά, στα χωρικά μας ύδατα, στα νησιά Συνκάκου. Παραβίαση των υδάτων. Αυτό αποτελεί πρόκληση. Και επίσης έχουμε και εκφοβισμό. Πολύ σημαντικό και αυτό το φαινόμενο. Και αφορά όλη την περιοχή. Τέλος, για τα περιφερειακά ζητήματα, να περάσω στη διαφάνεια 14. Όταν μιλάμε για Ανατολική Ασία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και τη Ρωσία είναι και αυτή γείτονε μας. Και δικό σα και δικό μας και δικός μας. Έχουν παραβιάσει και το εναέριο χώρου μας ε, και οι αναχαιτήσεις είναι σχεδόν ε, καθημερινό φαινόμενο. Τέλος 15 σελίδα. Και έχουμε και πολλές παρεμβολές. Στη σελίδα λοιπόν 15 τώρα όπως ε, έλεγα, η θάλασσα της Ανατολικής Κίνας μας δημιουργεί προβλήματα, αλλά Ε, θα έλεγα ότι υπάρχουν και αντιστοιχίες με το τι γίνεται με την Κρυμαία και την Ουκρανία. Διότι εδώ υπάρχει προσβολή ε, και αμφισβήτηση του στάτους κβό. Είτε δια της βίας είτε δια του εξαναγκασμού. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε και αυτό το είπε και ο Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιαπωνίας. Επιβλήθησαν κυρώσεις ε, στη Ρωσία για την Κρυμαία. Θα θέλαμε αντίστοιχα η ενεργή και δραστήρη να είναι οι Ευρωπαίοι φίλοι μας και σε σχέση με τα όσα γίνονται στην Ανατολική Ασία. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο ε, θέμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ σήμερα. Τι θέλει δηλαδή η Απωνία να πετύχει με τη νέα νομοθεσία για την ασφάλεια βασιζόμενοι στα όσα συμβαίνουν γύρω από την ε, Ιαπωνία, πέρασε μια καινούρια νομοθεσία για την ασφάλεια την ε, ε, προηγούμενη χρονιά, όπως εξήγησε και ο κύριος Πρέσβης. Θα με ρωτήσετε ποιες είναι οι αλλαγές που επιφέρονται. Θα σας πω ότι υπάρχουν τρεις κύριες αλλαγές. Πρώτον, ευρύτερη συμμετοχή της Ιαπωνίας στις διαδικασίες ειρήνευσης των Ηνωμένων Εθνών και άλλες ε, προσπάθειες ε, που την χάνουν διεθνού συντονισμού. Όπως, ε, υπεγράφει, όπως τονίστηκε και από τον πρέσβη Κατακάμι, εμείς προσεκτικά παρακολουθούμε τα όσα κάνει η Ευρώπη και όσα ε, ε, ε, τελούνται στα πλαίσια των αποστολών της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας ας πούμε η Ιαπωνία συμμετείχε στην διαδικασία, στην επιχείρηση Αταλάντη της NAVFOR. Δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η ενίσχυση της ηλικής ε, ε, ε, στήριξης της Ιαπωνίας σε άλλες αποστολές στο Αφγανιστάν, ας πούμε, επιχειρήσεις προς το Αφγανιστάν. Ε, μέσω αυτής της νομοθεσίας ε, θα έχουμε πλέον την νομική βάση έτσι ώστε η Ιαπωνία να μπορέσει ε, να συμβάλλει σε αναλώσιμα που δεν θα είναι πλέον απλώς ε, κάποια ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα κτλ, αλλά και συγκεκριμένη ε, συμβολή με προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Τρίτον, ε, τρίτο μεγάλο στοιχείο είναι η άσκηση του δικαιώματος συλλογικής αυτοάμυνας. Όλα τα έθνη, όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν την δυνατότητα της ατομικής αυτοάμυνας αλλά και της συλλογικής αυτοάμυνας. Λόγω της ερμηνείας του Ιαπωνικού συντάγματος εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα συλλογικής αυτοάμυνας μέχρι τώρα. Μέσω της νέας νομοθεσίας με περιορισμένο τρόπο θα έχουμε την δυνατότητα να ασκήσουμε το εν λόγω δικαίωμα. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτές δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ίσως ε, το πει κάποιος αυτό ε, ίσως αυτό αυτά που σας λέω να σας φαίνονται πολύ βασικά, ε, αλλά πρέπει να σας πω ότι για μας ε, οι αποτελούν μέγιστες ε, μίζωνες αλλαγές στο ιαπωνικό σύστημα ασφάλειας τα τελευταία 40 χρόνια, για να μην πω μετά τον πόλεμο. Μπορεί να είναι απλά, αλλά είναι πολύ βασικά. Τέλος, έχουμε και μία ενδιαφέρουσα σχημομέτρηση της κοινή γνώμης. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι λόγω αυτής της ε, νέας ε, νομοθεσίας ασφάλειας ε, και λόγω του ότι κάποιες φωνές αντίδρασης ακούστηκαν στην Ανατολική Ασία ε, ότι ίσως ο κόσμος ε, δεν ε, θέλει τις αλλαγές αυτές. Είναι μέγα σφάλμα, διότι η σιγομέτρηση αυτή καταδεικνύει ότι η Ιαπωνική κοινωνία δέχεται αυτές τις αλλαγές. Βέβαια, σε σχέση με την Κίνα ή με την Ρωσία ε, ε, πραγματικά βλέπει κανείς και διαπιστώνει ότι στην Ιαπωνία δεν θέλει ε, ο κόσμος στρατιωτικές λύσεις. Ίσως θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα, αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να σταματήσω εδώ έτσι ώστε να υποβάλλετε εσείς τα ερωτήματά σας. Okay, Πολύ ωραία. Παρακαλώ, αν έχετε ερωτήσεις. Ο κύριος Πασκού, παρακαλώ, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή και έχετε απόλυτα δίκιο. Είπατε κάποια στιγμή ότι μέχρι τώρα δεν σας επέτρεπα να κάνετε κάποια πράγματα που τώρα σας επιτρέπονται. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια αυτοεπιβαλόμενη πολιτική με την έννοια ότι εσείς είχατε αποφασίσει ότι δεν θα κάνατε κάποια πράγματα. Δεν είναι ότι κάποιος απ' έξω σας επέβαλε κάποια άλλα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι ότι υπάρχει μια διεθνή συμφωνία που τροποποιήθηκε, απλά είναι δική σας η απόφαση. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι στην Ευρώπη χαιρετίζουμε τη νέα σας πολιτική και τη διάθεσή σας να στηρίξετε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε διάφορες περιπτώσεις, θέατρα πολέμου ενδεχομένω. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι το βασικό μας πρόβλημα δεν είναι ότι μας λείπουν οι σύμμαχοι, αλλά μας λείπει η πολιτική βούληση μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Αν πάρουμε την περίπτωση στο Μαλί, θα δούμε ότι μόνο η Γαλλία είναι παρούσα στο Μαλί. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να λύσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα. Φαντάζομαι γνωρίζετε ότι θα χαιρετήσουμε οποιαδήποτε απόφαση της Ιαπωνίας να στηρίξει κάποιες επιχειρήσεις και υπάρχουν ε, πολλές ε, περιπτώσεις που χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Όμως ε, διαρωτώ και αυτό είναι ένα ερώτημα προς εσάς. Διερωτώ για το κατά πόσον η συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα ε, ναυτικής επίσης ή όχι, γιατί υπήρξαν κάποια θέματα επιμελητίας στα οποία συνεργαστήκαμε. Αρκεί αυτό έτσι ώστε η μελλοντική μας συνεργασία να αρχίσει να λειτουργεί ευθύς εξ αρχής ή μήπως ε, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να προσαρμοστείτε κι εσείς ε, στον τρόπο με τον οποίο εκτελούν οι Ευρωπαίοι κάποια παρεμφερή καθήκοντα ή αποστολές. Ο κύριος Γκάλα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε για τις νέες πολιτικές που θα ακολουθήσει η, η Ιαπωνία. Εγώ από τη Γερμανία και κατά τη διάρκεια των ετών είχαμε είτε περιορισμούς ε, που επιβάλλονται άμεσα από τους ε, συμμάχους μετά τον πόλεμο ή αυτοπεριορισμούς και μετά την ε, επανένωση στόχος ήταν να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, σε ένα κόσμο όπου δεν θα μπορούσε κανείς να κρυφτεί πίσω από τα, ε, τις παλιές συνήθειες του αυτοπερισμού. Έτσι λοιπόν μπορώ να φανταστώ ότι και στη δική μας τη χώρα έγιναν παρεμφερείς ε, συζητήσεις και τα έχετε ακούσει αυτά. Αυτή η ενέργεια της ε, κυβέρνησης δεν έγινε με ευρεία συνένεση και ρωτώ υπάρχει στο Κοινοβούλιο ή γενικότερα ε, κάποια συζήτηση με εμπειρογνώμονες, με κόμματα για το πώς είναι δυνατόν να διευρυνθεί πολιτικά αυτή η προσέγγιση. Έτσι ώστε να μην προκύπτει μια κατάσταση όπου όταν αλλάζει κυβέρνηση να επαναρχόμαστε στο σημείο 0. Δηλαδή τι θέλω να πω, να πιστούν περισσότεροι για την επιστροφή στην κανονικότητα. Ε, τι γίνεται σχετικά με αυτή τη συζήτηση. Αυτό ήθελα να μάθω. Η κυρία Λούζινγκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ συνεχίζω εκεί που το άφησε ο συνάδελφός μου αυτά που μόλις τώρα είπε ο συνάδελφος κύριος Γκάλα. Είπατε ότι τώρα μπορείτε στην Ιαπωνία να κάνετε πράγματα που δεν μπορούσατε να κάνετε στο παρελθόν και αυτό έγινε με απόφαση της κυβέρνηση. Το ερώτημα που τίθεται βέβαια είναι κατά πόσον αυτή η αλλαγή κατά πόσον αυτή η απόφαση κυβέρνηση ε, είναι συνταγματική ή όχι. Γιατί ξέρετε, με... μου κάνει εντύπωση το ότι μπορεί να υπάρξει, γίνεται αυτή η αλλαγή, παρότι ο κύριος Γκάλε αυτή την αλλαγή τη χαρακτήρισε ως ε, κανονικότητα. Ίσως και το παλαιότερο να ήταν το κανονικό. Είναι ένα θέμα αυτό. Πάντως, στο άρθρο 9 του συντάγματός σας ε, αναφέρεται αυτός ο προσανατολισμός. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ και εγώ πώς είναι δυνατόν παρά την ε, κατοχήρωση ε, στο Σύνταγμα να λέτε ότι τώρα είναι δυνατό κάτι που δεν ήταν δυνατό κατά το παρελθόν. Μήπως αποσκοπείτε σε συνταγματική αναθεώρηση. Αν ναι, τότε αυτό ε, κατευθύνεται προς αυτό που είπε ο κ. Γκάλερ. Τι θα γίνει δηλαδή αν ε, μελλοντικέ κυβερνήσεις είναι άλλη γνώμη, μήπως ε, αποσκοπείται σε συνταγματική αναθεώρηση. Και μία άλλη ερώτηση. Μιλήσατε για την κατανόηση από πλευράς κοινή γνώμης η οποία πρέπει να αποκτηθεί ακόμα σχετικά με τις αλλαγές που έλαβαν χώρα. Μερικές φορές το θέμα δεν είναι μόνο της ε, διαμεσολάβησης, ε, τα στατιστικά δεδομένα το δείχνουν αυτό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η άποψη στους ε, πολίτες και στη Γερμανία ισχύει το ίδιο. Δηλαδή οι πολίτες δεν συμφωνούν πάντα με αυτά που κάνουν οι κυβερνήσεις. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία οι σφιγομετρήσεις δείχνουν ότι 80% των πολιτών τάσεται κατά της Τη συμμετοχή στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Η κυβέρνηση βέβαια αποφάσισε διαφορετικά, τώρα δεν θα το συζητήσουμε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη δική σα τη χώρα το θέμα δεν είναι ακαδημαϊκή φύση. Διάβασα ότι αυτή τη στιγμή ο Οκινάβα, στην Οκινάβα μάλλον, διαφωνεί ο διοικητή, Διαφωνεί στην περιοχή αυτή, στην Οκινάβα, να ε, υπάρξει αμερικανική στρατιωτική βάση. Και το θέμα δεν είναι απλά αντικείμενο συζητήσεων. Αυτή τη στιγμή είναι ε, αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις σε αυτή την αλλαγή. Ο εν λόγω διοικητής εξελέγει ακριβώς διότι στήριξε την ειρηνευτική άποψη και ο ίδιος επίσης είχε καταφερθεί κατά της ε, στρατιωτικής βάσης. Γι' αυτό τον εξέλεξαν οι πολίτες. Άρα δηλαδή όλα αυτά μήπως δείχνουν ότι υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και άλλες περιοχές της Ιαπωνίας. Και ερωτώ κατά την άποψή σας τι θα γίνει στο μέλλον και έχω και μία άλλη συγκεκριμένη ερώτηση. Μιλήσατε για τις αντιπαραθέσεις ε, στην ε, θάλασσα της Νότιας Κίνας ε, μας τα περιγράψατε ως ε, μια επίμαχη κατάσταση. Η δική σας η στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των ε, διαφωνιών ποια είναι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτά που μας είπατε. Δύο ημέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου ε, συναντήθηκα στην Πολωνία με τον ε, Ιάπωνα πρέσβη. Τότε ε, ήμουνα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και ήρθε ο πρέσβης για να μας πει ότι παρότι η Ιαπωνία είχε βάσει του συντάγματος σοβαρούς περιορισμούς, παρόλα αυτά η Ιαπωνία επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μία ε, διεθνή προσπάθεια για να ε, διευκολύνει την κατάσταση προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, ήθελε η Ιαπωνία να προσχωρήσει και αυτή τη Συμμαχία Αντιμετώπισης της ε, Τρομοκρατίας. Ήθελε να στείλει βοήθεια με πλοία, με ανθρωπιστική βοήθεια και το καθεξής. Από ό,τι είχα δηλαδή καταλάβει, ήταν το πρώτο βήμα που θα οδηγούσε σε αυτό που υπάρχει σήμερα κατά κάποιον τρόπο. Επιπλέον, η συμμετοχή σας ε, στην Ουκρανία, ούτε και αυτό είναι κάτι το καινούριο. Θυμάμαι περίπου την ίδια περίοδο ε, θυμάμαι τη συμμετοχή σας σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα και αργότερα ε, συμμετείχατε με διάφορους τρόπους ε, σε σχηματισμούς που ήθελαν να εμπλακούν στη διαμάχη στην Ουκρανία. Τώρα, στο Μαλί είσαστε παρόντες σε όλες ε, τις περιοχές που είναι πολύ σημαντικές ε, για θέματα ασφάλειας. Στην Αφρική βλέπουμε ότι αποσταθεροποιούνται σημαντικά κομμάτια της περιοχής. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Και το ίδιο ισχύει και για προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εξ ανατολών. Όλοι το ξέρουμε αυτό, ότι είναι απαραίτητο να στηρίξει κανείς την Ουκρανία έτσι ώστε η Ουκρανία να έχει μια σταθερή κυβέρνηση και να μπορεί να αντισταθεί σε όλες τις ε, προκλήσεις που μπορεί και να προκύψουν. Εγώ χαιρετίζω όλες αυτές τις εξελίξεις για συνεργασία ε, και σε επίπεδο ασφάλειας και άμυνας. Τελικά Ίσως αυτά χρειάζονται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών θα δούμε κατά πόσον ε, μπορούμε να εξετάσουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Όσον αφορά στην ύπαρξη πυρηνικών δυνάμεων γύρω από την Ιαπωνία και αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Ε, πράγματι φαντάζομαι κάτι έχετε διαπιστώσει, ε, κάτι το οποίο έχει ήδη αναφερθεί και γι' αυτό το λόγο αποφασίσατε να είστε λίγο πιο ε, κατηγορηματικοί όσον αφορά τα αμυντικά σας σχέδια τα κατανοούμε αυτά και ευχόμαστε τα καλύτερα για σας και για το λαό της, της Ιαπωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τις ερωτήσεις. Τις θεωρώ όλες πολύ σημαντικές. Πρώτα απ' όλα, να αναφέρω πολύ ξεκάθαρα ότι η Ιαπωνία είναι μια δημοκρατική χώρα είναι σταθερή ε, δημοκρατία. Άρα είναι φυσικό να υπάρχουν στην Ιαπωνία πολλές διαφορετικές απόψεις σε σχέση με την νέα νομοθεσία περί ασφάλειας. Στη σελίδα 25 εξηγώ ότι είχαμε πάρα πολύ ενδελεχείς συζητήσει για την νομοθεσία αυτή. Εφτά χρόνια συγκεκριμένα κράτησαν οι συζητήσεις ε, το πάνελ των εμπειρογνωμόνων και έπειτα είχαμε και στην Ιαπωνική Βουλή μία πάρα πολύ αναλυτική συζήτηση. Αλλά ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε και να αναλάβουμε δράση. Ίσως λοιπόν να υπάρχουν κάποιες φωνές που εκφράζουν κάποια αντίθεση ε, η αντίδραση, αλλά αυτό είναι δημοκρατία. Ελήφθη η απόφαση πάντως και η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τώρα αυτή την απόφαση. Σε ό,τι την πρώτη ερώτηση. Σίγουρα απαιτείται προετοιμασία. Η κυβέρνησή μας, ε, κατά την άποψή μου, ε, επιδεικνύει επαρκή ε, προ, επαρκή σύνεση και σοφροσύνη και προχωρά με πολύ προσεκτικά βήματα. Δεν θα ληφθούν βιαστικές αποφάσεις, ιδίως όταν αυτές αφορούν και απαιτούν ε, την ανάληψη τακτικής δράσης. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε προώθημοι και διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε ακόμη περισσότερο στη διεθνή ειρήνη και επιμέρεια Η συμμετοχή λοιπόν στις ειρηνευτικές ε, επιχειρήσεις του ΟΗΕ θα είναι πολύ πιο ομαλή από ό,τι πιο πριν. Αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση. Σε ό,τι αφορά τώρα κάποια άρθρα, το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 9 του Συντάγματος της χώρας μου προβλέπει ότι η Απονία απαρνείται τη χρήση βίας ή ε, την απειλή της χρήσης της βίας ως τρόπο επίλυσης των διεθνών διαφορών και διανέξεων. Και μέχρι εκεί σταματάει. Δεν προβαίνει σε καμία ειδική αναφορά είτε στην ατομική είτε στη συλλογική άμυνα. Όμως, η αυστηρή μήνυ αυτού του άρθρου υπερτερούσε μέχρι τώρα από την έννοια αναφορα ειτε στην ατομικη ειτε στη συλλογικη αμυνα ομως η αυστηρη αυτου του αρθρου υπερτερουσε μεχρι τωρα με την εννοια οτι όπως προβλέπει αυτό το άρθρο, η Ιαπωνία απαγορεύεται να καταφύγει σε μέτρα ε, συλλογικής άμυνας. Όμως υπάρχουν άλλα διατάξεις. Πάνω χάρη, το προήμιο του Ιαπωνικού Συντάγματος τονίζει τη συμβολή της Ιαπωνίας στην ε, διεθνή κοινότητα. Γιατί λοιπόν να κάνει παραπάνω η Ιαπωνία. Γίνονται συζητήσεις, ακούγονται επιχειρήματα, δυνάμει της νέας ερμηνείας του ίδιου συντάγματος αποφασίσαμε όχι μόνο ε, ατομικό το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αλλά το δικαίωμα και στη συλλογική αυτοάμυνα να επιτρέπεται. Αυτή την απόφαση την πήρε η Βουλή. Ήταν μια δημοκρατική διαδικασία, διαφανής διαδικασία, και όπως προείπα προηγήθηκαν εντελεχέστατες συζητήσεις. Ναι, ο κυβερνήτης της Οκινάου έχει κάποιες περίεργες ιδέες σε ό,τι αφορά τη συμμαχία Ιαπωνίας Ιαπωνίας-ΕΠΑ Πολιτειών. Αλλά αναφέρει και το λέω και εγώ, ότι υπάρχουν και στην Οκινάουα διαφορές και ε, στις απόψεις. Εμείς προχωρούμε πολύ προσεκτικά, λαμβάνουμε υπόψη τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται στην Οκινάουα και προσπαθούμε να καταλάβουμε καλύτερα και την τοπική κοινωνία και την ανάγκη να ενισχύσουμε την συμμαχία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, ποια είναι η στρατηγική μας για τη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Ε, θα σας δώσω μια απλή απάντηση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πολυμερές σύστημα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα και τους μηχανισμούς της ειρηνικής επίλυσης διαφορών. Και η κυβέρνηση των Φιλιππίνων έκανε προσπάθεια να φέρει το ζήτημα σε διεθνή διαιτησία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρετηθεί και να επικροτηθεί αυτή η προσπάθεια από οποιαδήποτε χώρα υποστηρίζει το κράτος δικαίου. Το να στέλνετε τα πλοία σας σε αμφισβητούμενα είδατα δεν βοηθάει να λυθούν. Ούτε οι εκφοβισμοί, ούτε ο ξαναγκασμός βοηθάει. Ζούμε σε μια κοινωνία που βασίζεται σε κανόνες. Γιατί λοιπόν να μην καταφύγουμε σε ένα μηχανισμό που είναι διεθνώς ε, και νομικά κατοχυρωμένος. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σύντομη απάντηση που μπορώ να σας δώσω σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά περιεκτική παρουσία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, και εσάς, κύριε Γενική Διευθυντά, γιατί μας ενημερώσατε με πληρέστατο τρόπο για τι πρόσφατες αλλαγέ, στην νομοθεσία περί ειρήνη και ασφάλεια στην Ιαπωνία. Σας ευχαριστώ θερμά. we can immediately transfer to the next point of our agenda. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης. Και συγκεκριμένα θα εξετάσουμε την ε, έκθεση Van Orden. Πρόκειται για μια έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας θέμα της έκτασης ιδέας πρωτοβουλίας είναι οι υπηρεσίες υποστήριξης της ειρήνης ε, και η ε, συμμετοχή της ΕΕ σε συνεργασία με τα ΗΕ και την Αφρικανική Ένωση. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για τη δέσμευση που έχει αναλάβει λοιπόν ΕΕ με ΝΑΤΟ και Αφρικανική Ένωση λίγη προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 23 Φεβρουαρίου, θα συζητήσουμε το Μάρτιο για δεύτερη φορά την έκθεση και τον Απρίλιο. Α, στην ΑΦΕΤ πρώτα, ναι, και μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Κύριε Βανόρντεν, Μπορείτε να μας παρουσιάσετε τις βασικές ιδέες της έκθεσής σας. Πρώτα απ' όλα, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί η βοήθειά σας. Ήταν πάρα πολύ πολύτιμη στο να ε, συντάξω αυτή την έκθεση και επίσης να ευχαριστήσω και τον επικεφαλής του συνδέσμου, γραφείου συνδέσμου στις Βρυξέλλες, γραφείου συνδέσμου των Ηνωμένων Αθνών, ε, γιατί προσέφερε την υποστήριξή του ε, για αυτή την έκθεση. Η ουσία τώρα που στοχεύει η έκθεση είναι το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποδώσει υπεραξία ε, και βλέπουμε το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις δραστηριότητες και πολλών άλλων. Ε, το κυριότερο αφορά την ε, ε, Αφρική. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι θα πρέπει κάπως να, να, να, να φανεί αυτό στον ε, τίτλο. Εγώ θα προτιμούσα βεβαίως ο, ο τίτλος να είναι ε, ε, οι επιχειρήσεις υποστήριξης στην Αφρική. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω δεν ε, γίνεται γιατί βλέπω ότι κουνάτε το κεφάλι σας αρνητικά. Εν πάση περιπτώσει. Εθνικές κυβερνήσεις, ε, πολυεθνικοί οργανισμοί κτλ. Ε, όλοι όσοι ασχολούμαστε χρόνια με την Αφρική είναι να αυξηθεί η ικανότητα ε, που θα έχει για να λύσει τα προβλήματα της Υπήρου. Επομένως είναι ζωτική σημασία οποιαδήποτε δέσμευση προς την Αφρική να αφορά κυρίως την οικοδόμηση ικανοτήτων. Και αυτό άλλωστε είναι και ο μύθος της αδιάγνησης σε αυτήν την ε, έκθεση. Ε, η διαδικασία ε, δυνατότητας ε, ε, επιχειρήσεων, από αυτήν την ε, δύναμη υποστήριξης της ειρήνης βασίζεται βεβαίως και η αναδιπλώσή της, η, συγγνώμη, η ανάπτυξή της βεβαίως εξαρτάται και από την καλή βούληση των ιδίων. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι και βεβαίως εδώ τα μάλλα μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως χρειάζεται ε, μεγαλύτερη ε, απόδοση ε, ευθυνών, οπωσδήποτε χρειάζεται... Uh, this obviously is also ε, Οπωσδήποτε χρειάζεται μεγαλύτερη ε, λογοδοσία και ε, φυσικά εμείς θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούνται καλά και δεν υπάρχει διασπάθηση των πόρων που προωθούνται προς τα εκεί. Βεβαίως εμείς δεν είμαστε οι μόνοι οι οποίοι καλούμεθα να διορθώσουμε όλα τα λάθη του κόσμου. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δεσμεύονται ε, μαζί με μας. Επομένως, ε, καλή και αποτελεσματική επικοινωνία ε, προς μεταξύ όλων αυτών των φορέων προς αποφυγή επικαλύψεων είναι ζωτική σημασίας. Εδώ βεβαίως θα πρέπει να αναφέρουμε και την ανάγκη αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Αφρική που είναι μια μεγάλη πληγή και η οποία αντιμετώπιση είναι ουσιώδους, θεμελιώδους σημασίας έτσι ώστε να γίνει αποτελεσματική η οποιαδήποτε ε, επιχείρηση. Ελπίζω να διαπίστωσαν ήδη οι συνάδελφοι ότι πολλές από τις παρατηρήσεις τους έχουν ήδη ενσωματωθεί στην ε, έκθεση και βεβαίως ε, σημαντικό είναι να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο και ε, βεβαίω πρέπει να ε, περιληφθούν όσο γίνεται περισσότερα στην έκθεση έτσι ώστε να είναι λίγες οι τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις ε, εισηγητές γιατί βλέπω ότι αρκετοί μεταξύ αυτών είναι εδώ. Θα δώσω ας πούμε πρώτα απ' όλα τον λόγο στον κύριο Ζηρίσκη εξ του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Έχουμε χρόνο. Αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν θα μιλήσω ε, πολύ. Πρόκειται εδώ για μια έκθεση η οποία είναι συγκεκριμένη, είναι συνοπτική, αναφέρεται ε, σε ε, λύσεις. Έχουμε ας πούμε την σύσταση για αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και σωστή επικοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο κύριος Βανόρντεν τα έχει πολύ καλά αναφέρει. Ίσως ε, καλό θα ήταν να προσθέσουμε δύο στοιχεία. Πρώτον, για να υπογραμμίσουμε την ε, εκπαίδευση και την ε, κατάρτιση έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη χρήση των πληροφοριών do pokazania przykładu kompleksowego radzenia sobie. Και e, επειδή ακριβώς e, e, θα πρέπει να, να μάθουμε στους ενεχομένους και εμπλεκομένους τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επιλύουν ε, τις ε, διαφωνίες. Και κάτι άλλο. Το πί και το R, τα δύο αυτά θέματα ε, έχουν κάποια στοιχεία επί των οποίων είχαμε συμφωνήσει από την αρχή γιατί είχαμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν θα πρέπει να επικαλύψει ε, εργασία άλλων. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει για δεύτερη φορά κάτι που κάνουν άλλοι. Να δούμε λοιπόν μήπως το θέμα αυτό να είναι ας πούμε κρίσιμο. Στο άρα επίσης αναφέρεται ότι ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι θεσμικές ε, προτάσεις ε, και αναφέρεται ότι ενδεχομένως μεγαλύτερες φιλοδοξίες να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Εγώ δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μία διατύπωση διαφορετική έτσι ώστε το κείμενο να γίνει πιο σαφές και να μην υπάρξει καμία εύλογη αμφιβολία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζιλ Περνιέ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον Τζέφρι Βαν Όρντεν, για την εξαιρετική και ποιοτική εργασία του, αλλά και για τον επαγγελματισμό του. Το θέμα που μας απασχολεί εδώ ε, είναι φλέγον. Το θέμα της ε, ασφάλειας στην Αφρική, κυρίως δε στην περιοχή του Σαχέλ, δηλαδή ε, πρώτων πυλών της Ευρώπης, είναι κάτι που μας απασχολεί. Έχουμε τη Σεμπάμπ, έχουμε την Μπόκο Χαράμ, έχουμε στο Μαλί, στον Νίγηρα, στην Πουρκίνα, Φάσο, ένα σωρό οργανώσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα καθημερινά. Βεβαίως ε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι επιτόπου, εργάζονται μαζί με άλλους εκπροσώπους διεθνών οργανισμών έτσι ώστε ε, μαζί με τους Αφρικανούς, μαζί με την Αφρικανική Ένωση και με τα Ηνωμένα Έθνη να ξεκινήσουν διαδικασίες οι οποίες εν τέλει θα ωφελήσουν από πλευράς ασφάλειας ε, την ίδια την Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό είναι και η ουσία και το συμπέρασμα του, ε, της έκθεσης Βανόρντεν. Ε, να πω δύο λόγια λοιπόν. Πρώτα απ' όλα αγαπητέ συνάδελφε, σας στηρίζουμε απολύτως για την προτεραιότητα που θέλετε να δώσετε στις αφρικανικές δυνάμεις. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε τους Αφρικανούς έτσι ώστε μόνοι τους να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Η βοήθειά μας θα πρέπει να εστιαστεί περισσότερο σε διαρθρωτικές χρηματοδοτήσεις όπως είναι η κατάρτιση ή ε, ο εξοπλισμός ε, και οι πόροι να διασπαρούν σωστά σε ολόκληρη την, ε, την Αφρικανική Ήπειρο. Αυτή τη στιγμή περισσότερες χρηματοδοτήσεις δίνονται στη Σομαλία και 80% χρησιμοποιείται έτσι ώστε να πληρωθούν οι μισθοί των στρατιωτών. Ενώ πλέον ξέρουμε ότι ήδη στο νότο του, της Λιβύης, ήδη ένα σωρό άλλες γεωγραφικές περιοχές έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω ακριβώς των τρομοκρατικών οργανώσεων που εκεί λειτουργούν και επομένως θα πρέπει η χρηματοδότηση ε, να διαρθρωθεί διαφορετικά και να ε, στηριχτούν οι ικανότητες και οι δυνατότητες των Αφρικανικών στρατών. Επίσης, ε, ε, πέραν της ε, ήδη καλής παρουσίας της Αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολλές δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης. Ας πούμε, η δυνατότητα αξιολόγησης πριν και μετά των στρατιωτικών δυνάμεων. Δεύτερον, θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή παρέμβαση δεν θα πρέπει να γίνεται μονάχα από αποστολές PSDC επιτόπου να συνεχίσουμε ε, ε, ε, γιατί να συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάποιες δυνάμεις γιατί ας πούμε οι δυνάμεις της Γαλλίας επιτόπου δεν προσπαθούν να διασφαλίσουν τα γαλλικά συμφέροντα αλλά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και επίσης δεν θα πρέπει να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ενοχλεί, να παρενοχλεί την εργασία άλλων οργανισμών επιτόπου, αλλά θα πρέπει να συμβάλλει γιατί στην παράγραφο 12, αυτή η ιδέα είναι παρούσα λίγο, στην παράγραφο 12 της εργασίας του κυρίου ε, Βαν Όρντεν. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ε, αναφέρουμε ότι πιο συστηματικά θα πρέπει να αναφέρονται οι προσπάθειες. Επίσης, Ε, θα πρέπει οι ε, περισσότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις να ακολουθήσουν ε, την ενεργοποίηση του άρθρου 42-7 <clears throat> από τη Γαλλία. Τέλος, κάτι το οποίο θα θέλαμε πιο πολύ να εμφανίζεται στην έκθεση είναι η συνεργασία με, τις άλλες, με τους άλλους οργανισμούς, κυρίως όσον αφορά τους, τα, τα σύνορα. Αυτό αναφέρεται ήδη ε, ε, ήδη στην αιτιολογική σκέψη C, βεβαίως το πορότες των συνόρων είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ε, και αφορά όλη την περιοχή του Σαχέλ. Κατά την άποψή μου αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι ένα, ένας από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής επένδυσης ας πούμε σε αυτήν την επιχείρηση. Αυτά είναι κυρία Πρόεδρε οι γενικές γραμμές επί των οποίων θα βασιστούν οι τροπολογίες μας και πριν τελειώσω να συγχαρώ τον συνάδελφο Όρντεν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Περνιό. Ο κύριος Φανάρτ ε, είναι ο σκιώδης ε, ε, εισηγητής για την Άλντε, αλλά λείπει και επομένως θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ράντος να μας πει, την, να κάνει την παρέμβασή του όσον αφορά το θέμα του κύριου Βανόρτ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Ξαβιέ Νάρτος και ο δισηγητής της πολιτικής ομάδας ε, δεν μπόρεσε να έρθει γιατί συμμετέχει στην αντιπροσωπεία του ΕΛΚ ε, για την παρατήρηση εκλογών στην Ουγγάντα και μου ζήτησε με λίγα λόγια να εξηγήσω, να παρουσιάσω τη θέση του ε, σε, αυτή το, σε αυτό το σχέδιο έκθεση. Ευχαριστεί λοιπόν ο συνάδελφο, τον κύριο Βανόρντεν, για αυτό το σχέδιο έκθεση. Επίση και για τι προσπάθειε που κατέβαλε ευθύ εξ αρχή να επιτευχθεί η συνένεση. Ο κύριο Νάτα συμφωνεί με αυτό το σχέδιο έκθεσης, ε, θεωρεί ότι είναι πολύ ακριβής ε, και λογική. Υπάρχουν όμως δύο βασικά θέματα όπου ο κύριος Νάτα ε, θεωρεί ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση του κύριου Βανόρντεν. Και γι' αυτό το λόγο θα καταθέσει τροπολογίες. Πρώτον, να αναφέρεται το γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση κατάφορης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η τρομοκρατική απειλή απειλούν την ειρήνη και τις αποστολές ε, αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση γιατί η ειρήνη δεν μπορεί να διαφυλαχθεί αν καταρχήν δεν έχει επιτευχθεί. Τον δεύτερο ε, αναφέρεται η αναγκαιότητα να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα από όλα τα μέλη των ειρηνευτικών αποστολών και να υπάρχει μια στρογγυλή τράπεζα για αυτά τα θέματα. Οι χώρες που αποστέλουν στρατεύματα στις ειρηνευτικές αποστολές ε, δεν ε, δέχονται και δεν σέβονται όλες αυτές οι χώρες τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς όμως ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ε, βασικός ιδρυτής αυτών των αποστολών πρέπει να διασφαλίζουμε την, ε, την, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως και ο δισηγητής της ομάδας των φιλελευθέρων επιθυμεί να υπογραμμίσει την υποστήριξή του προς αυτό το σχέδιο έκθεση. ευχαριστούμε πολύ. Και... Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Κόζο Περμούη δεν θα παρέμβει. Ε, επομένως θα δώσω το λόγο στην κυρία Μποντίλ Βαλέρο από του Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ, λυπούμε πολύ που άργησα και δεν άκουσα από την αρχή γιατί ήμουν σε μια άλλη επιτροπή. Ξέρετε πώς δουλεύουμε σε αυτό το σώμα. Ήταν πολύ καλή βιβλία του κ. Βανόρντεν ήδη και βλέπω ότι κάποιες από τις δικές μας ε, συστάσεις έχουν ε, περιληφθεί στο κείμενο στην ομάδα μας. Ε, συζητήσαμε το ενδεχόμενο να προσθέσουμε κάτι περισσότερο για τα οικονομικά για τη χρηματοδότηση. Πάτε στην αρχή θα πρέπει να γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Το 2003 όμως αυτό ισχύει και θα πρέπει να είναι προσωρινό. Άρα θα υποβάλουμε σχετικέ τροπολογίες. Σε ό,τι διάφορα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Είδαμε σε διάφορες αποστολές το πρόβλημα στην κεντροαφρικανική δημοκρατία και σε άλλες χώρες παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Το είδαμε και όχι εμείς μόνο και σε αποστολές το ΟΗΕ παρατηρείται και συνεχώς καταγράφεται και πρέπει να το αναφέρουμε στην έκθεση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μικαλ Γκάλερ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ τα ήθελα να συμφωνήσω με τη θετική αξιολόγηση της έκθεσης. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος στο Γεύσκι αλλά και ο συνάδελφος Πανιό. Ε, συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε ε, να ε, ενισχυθεί η ίδια πρωτοβουλία για την ειρήνη στην Αφρική. Δηλαδή, όχι εμείς να προσφέρουμε απλά ειρηνευτικές αποστολές και να βασίζεται σε αυτές η Αφρικανική Ένωση. Η ίδια η Αφρική ε, θα πρέπει να συμμετέχει στο οικοδόμημα για την ειρήνη και στις εφεδρικές δυνάμεις. Εκεί να επιδείξουν την πολιτική βούληση να αναλάβουν δράση στην ε, συνεδρίαση ασφαλείας που έλαβε χώρα στο Μόναχο ε, συζητήθηκαν όλα αυτά τα θέματα σε ομάδες εργασίας. Ε, το πρόβλημα λοιπόν είναι γνωστό. Εγώ σκέφτομαι το κατά πόσον θα έπρεπε να συμβουλεύσουμε αυτές οι εχθρικές δυνάμεις ίσως να εγκατασταθούν στις περιφερειακές οργανώσεις γιατί η Αφρική είναι τόσο μεγάλη σε έκταση έτσι ώστε στο Σαχέλ ας πούμε ε, κανείς δεν νιώθει ότι είναι υπεύθυνο για το τι συμβαίνει στο βορρά της Αφρικής ή στους ωκεανούς είτε γίνει αυτό στο ΕΚΟΜΠΑ, στο ΙΓΑΤ ή στην East African ε, Community ή στη ΖΑΝΤΕΚ δεν έχει σημασία ε, η γεωγραφική ε, απόσταση παίζει ρόλο. Οι Αμερικανοί λένε ότι έχουν ένα πρόγραμμα ε, με βάση το οποίο οι ίδιοι ε, θα διαθέσουν το 75% των πόρων και οι Αφρικανοί μόνο το 25%. Αυτό μπορεί να με βοηθάει τώρα, βραχυπρόθεσμα, αλλά ε, θα πρέπει, όπως σας είπα παρόλα αυτά, να ενισχυθεί η λήψη ίδιας πρωτοβουλίας από πλευράς Αφρικανών. Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Φαντάζομαι τις περιμένει ο Τζόφρι από πλευράς μου. Ο συνάδελφος προηγουμένως αναφέρθηκε στο άρθρο 41 παράγραφος 2 όπου γίνεται λόγος για απαγόρευση στρατιωτικών δαπανών. Αυτό όμως αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, τις operations. Η δική μου η ερμηνεία είναι ότι πριν ή μετά μια συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί κανείς ε, να δαπανά πόρους. Και σημείο 13, παράγραφος 13, το περιμέναμε αυτό, αναφέρεται στα πολιτικά μέσα, μη στρατιωτικά δηλαδή, με αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα πρόγραμμα Train and Equip αν θυμάμαι καλά και αυτό το Equip, ο εξοπλισμός ε, εκεί τίθεται το ερώτημα κατά πόσον ε, κατά περίπτωση ε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στρατιωτικός εξοπλισμός για να υπάρχει λοιπόν μια ε, σφαιρική προσέγγιση. Ίσως ε, πρέπει, όπως σας είπα, να εντάξουμε στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα ε, για την αντιμετώπιση κρίσεων. Αυτά είχα να παρατηρήσω και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βανόρ δεν θέλει να σχολιάσει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους Κιώδης για την συνεχή τους ε, υποστήριξη. Οι παρατηρήσεις τους είναι θετικέ. Σε ό,τι αφορά τις παραγράφους P και R που αναφέρατε, θα τις απεξεργαστώ, αλλά νομίζω ότι όχι, δεν πρέπει να υπερβάλλουμε γιατί έχουν ε, κάποια φόρτιση και κάποια σημασία που αν αλλάξουμε και διατύπωση που μπορεί να χαθεί. Γι' αυτό ζητώ την κατανόηση των συναδέλφων. Τώρα, ναι, όλο αυτό το θέμα της ε, εφεδρικής ε, δύναμης από το Αφγανιστάν. Ε, πολύ σωστά τα είπε ο συνάδελφος Μίχαλε. Αν καταφέρουν περιφερειακές ομάδες σαν αυτή να τις κάνουν επιχειρησιακές θα είναι καλύτερα και σίγουρα πρέπει να το δούμε σοβαρά γιατί μπορούμε να τα συζητάμε όλα αλλά πρέπει να έχουμε και την εικόνα της πραγματικότητας γιατί θέλουμε μια δύναμη που να μπορεί να κάνει τη δουλειά της και να έχει έτσι περισσότερη ισχύει, περισσότερη εκπαίδευση, εξοπλισμό, οικονομική υποστήριξη και όλα αυτά. Και εμείς πρέπει να κάνουμε και τη δική μας δουλειά στις ε, πρωτεύουσες στις αφρικανικές, ε, να ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν, γιατί είναι σίγουρα και προς το δικό του συμφέρον. Δεν θα πούμε εμείς ποιο είναι το συμφέρον τους. Εμένα μου λένε ότι ναι, θέλουμε να το κάνουμε, απλά δεν ξέρουμε πώς. Αυτά είχα να πω, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα τι είπαν οι συνάδελφοι. Και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με επιτυχία. Πρόεδρος, θα σας υποσχεθώ και σε εσά και στους άλλους συναδέλφους ότι θα δω πολύ προσεκτικά τι μπορούμε να κάνουμε για να μην αλλάξει το θέμα αυτής της έκθεσης ιδίως πρωτοβουλίας. Ίσως να είναι δύσκολο ε, στην ε, πράξη, αλλά θα, θα σας ενημερώσω αν μπορούμε να αλλάξουμε το, το αντικείμενο. Εδώ ολοκληρώνεται η απογευματινή μας συνεδρίαση, αλλά ε, όπως με διορθώνουν, ξέχασα να σας πω ε, την προθεσμή κατάσταση τροπολογιών. 23 Φεβρουαρίου. 12 το μισή. Σας ευχαριστώ. Αύριο έχουμε πάλι πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Θα σας περιμένω. Καλό βράδυ.